Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην περιμένουμε περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλη η ημερήσια διάταξη μας, πάρα πολύ φορτωμένη. Όσοι δεν έχουν έρθει, τι να κάνουμε, θα χάσουν την ευκαιρία να ακούσουν τη σημαντική μας ενημέρωση. Αρχίζω για τις αποφάσεις των συντονιστών να σας πω ότι αποφάσισαν χθε οι συντονιστές. Δώσαμε εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις για τις νομοθετικές εκθέσεις, τις τεχνικές την τεχνική έκθεση την ανέλαβε ο ή πρόεδρος και το άλλο για την ετήσια ε, ποσόστοση για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης, δεν θυμάμαι πώς το λένε ακριβώς, ε, τον αναλαμβάνει η ε, ΓΚΟΕ για τις νομοθετικές γνωμοδοτήσεις. Επίσης η ΓΚΟΕ ζήτησε τη γνωμοδότηση για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Οι φιλελεύθεροι πήραν την έκθεση, μάλλον τη γνωμοδότηση για τη βιοπικιλότητα, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο ε, οι σοσιαλιστές, το μέλλον των αεροδρομίων οι φιλελεύθεροι, απαλλαγή 2010 το ΕΛΚ και επίσης αποφασίσαμε για τον τίτλο 3 ε, για τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Μία θα κάνει το ΕΛΚ για τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού ε, οι σοσιαλιστές θα πάρουν ε, για άλλη και για τη συνοχή για την Ευρώπη του 2020 πάλι σοσιαλιστές. Επίσης συζητήσαμε και συμφωνήσαμε για τις αντιπροσωπείες του 2012 τα ταξίδια της Επιτροπής στα γάλλο-ισπανικά σύνορα η πρώτη, η δεύτερη στην Κύπρο, η τρίτη στην Κοπεχάγη στα πλαίσια της Δανικής Προεδρίας. Επίσης συζητήσαμε για τις ακροάσεις και συμφωνήσαμε να κάνουμε τρεις μεγάλες δημόσιες ακροάσεις για το νομοθετικό πακέτο ε, για την πολιτική συνοχή και την Ευρώπη 2020 και τρίτη η πολιτική συνοχή και πώς ε, υποστηρίζει τις μακρόσιες επιχειρήσεις. Επίσης συμφωνήσαμε η επόμενη συνεδρίασή μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια του χρόνου να γίνει επίσης τον Οκτώβριο. Ξέρετε, σήμερα το απόγευμα ε, διεξάγεται και δεν ξέρουμε ακριβώς τα θέματα, αλλά θα συνδέονται με τα ε, νομοθετικά μέτρα, με τη δέσμη, αυτή τη νομοθετική. Ελπίζω να φτάνουμε τότε στο τέλος, στο διαπραγματεύσεο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε καλό είναι να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίσης, η ομάδα εργασίας για τη μελλοντική πολιτική συνοχής ε, θα συνεχίσει τις εργασίες της, όχι σε τακτή ε, βάση όπως σήμερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συζητούμε για την πολιτική συνοχή γενικότερα και πιο οργανωμένα. Ad hoc θα γίνει του χρόνου. Θα είναι γενικότερες οι ε, συνεδριάσεις και πιο δημόσιες, όχι μόνο για τους διαπραγματευτές ε, του νομοθετικού πλαισίου. Θα διατηρηθεί λοιπόν αυτή η ομάδα εργασίας και επίσης αποφασίσαμε για την επόμενη συνεδρία των συντονιστών που θα γίνει το Νοέμβριο να ετοιμάσει η Γραμματεία μια πρόταση και κατανομής ε, των πόντων ε, στις πολιτικές ομάδες για το δεύτερο ήμιση της θητείας. Αυτά. I would like to... Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη που είναι η εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρέχουσα πρακτική και μελλοντικέ προοπτικές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Ε, η συγκεκριτής είναι ο Φρανσουά Αλφόνση, ε, αλλά έχουμε και προσκεκλημένους ομιλητές, ε, στους οποίους θα ήθελα να δώσω το λόγο. Εξ ονόματο της Προεδρίας παρευρίσκεται η κυρία Ρίκα Μωσής Καντέντη, αναπληρώτρια διευθύντρια στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Πολιτικών στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας και ο κύριος Μπελάρτη από την περιφέρεια Μάρκε της Ιταλίας που είναι ειδικό και συνεργάζεται με τον εισηγητή στην ε, Επιτροπή Περιφερειών ε, για θέματα Αδριατικής ε, και Ιωνίων νήσου. Παρακαλώ, θα δώσω το λόγο στους ομιλητές μας για να μας ενημερώσουν πρώτα για τη Βαλτική, που είναι έτσι ένα μοντέλο που μπορούμε να υιοθετήσουμε και να ακολουθήσουμε για να έχουμε μια στρατηγική για την περιφερειακή πολιτική. Έχετε το λόγο παρακαλώ κυρία Μωσής Καντέντης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με χαρά βρίσκομαι ενώπιόν σας Έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις παρούσες ε, εξελίξεις και τις παρούσες συζητήσεις ε, σχετικά με την περιοχή της Βαλτικής. Για την Προεδρία είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό, διότι η στρατηγική για τη Βαλτική, επειδή είναι η πρώτη στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες είναι η υψηλότερη προτεραιότητα για το Συμβούλιο. Γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στη στιγμή που μετά από την πρώτη διετία εφαρμογής και υλοποίησης αναθεωρούμε τη στρατηγική αυτή για να δούμε ποια είναι τα πρώτα διδάγματα που αντλούμε, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και τι βελτιώσεις να κάνουμε. Η παρουσίαση μου διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Θα αρχίσω με κάποια βασικά στοιχεία για τη στρατηγική. Στη συνέχεια θα σας αναφέρω την πολωνική προσέγγιση και ε, τις βασικές παραδοχές, αν θέλετε, ε, για ε, τις διαδικασίες και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που βρίσκονται στο στάδιο της ε, προετοιμασίας. Ας αρχίσουμε λοιπόν με κάποια βασικά δεδομένα και γεγονότα. Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο ήταν εμπνευστή αυτής της στρατηγικής. Γι' αυτό χαίρομαι και πολύ περισσότερο που βρίσκομαι ενώπιον σας. Η στρατηγική για τη Βαλτική ε, και η ιδέα γεννήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006. By the Swedish Council. Uh, και το ε, ανέλαβε το 2009 η Σουηδική Προεδρία, όπου και εγκρίθηκε επίσημα και τυπικά βάσει της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε. Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική άρχισε να εφαρμόζεται εκκινώντας από την ιδέα να υπάρξει μια πρώτη θεώρηση ε, μετά από μια διετία. Όπως σας είπα, ακριβώς ε, μέσα του 2011 ε, κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τι κάνουμε Κάνουμε αναθεώρηση έτσι, όχι αξιολόγηση αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αξιολόγηση των ε, στρατηγικών αυτών των μακροπεριφερειών που είναι δύο ε, για τη Βαλτική και για το Δούναβη, θα γίνει το 2013, δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής. Ε, Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Τι είναι αυτή η στρατηγική. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική που καλύπτει διάφορα πεδία πολιτικής ε, της Ένωσης. Ε, πολιτική συνοχής, γεωργική πολιτική, υποδομές, μεταφορές κτλ. Και στοχεύει στη μακροπεριφέρεια όπως είναι η Βαλτική θάλασσα και όπως ορίζεται. Τέσσερις είναι οι πυλώνες και μπορείτε να τους δείτε στη παρουσίασή μου. Ο πρώτος είναι το περιβάλλον, ο δεύτερος η ευημερία, τρίτος ελκυστικότητα και προσβασιμότητα και το τέταρτο ασφάλεια ενεργητική και παθητική. 15 είναι οι τομείς προτεραιοτήτων. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια, το καθένα για διάφορες προτεραιότητες. Στην Πολωνία, ας πούμε, έχουμε δύο πολιτικές προτεραιότητες ή τομείς προτεραιότητας, το περιβάλλον κυρίως και η κατάσταση των υδάτων στη Βαλτική θάλασσα και τι γίνεται με τη ε, ρήπαση από τη Γεωργία. Και η δεύτερη προτεραιότητα που μας απασχολεί είναι η παριθμόν 7 που έχει να κάνει με την έρευνα και την καινοτομία. Είμαστε συναρμόδιοι και με ένα άλλο κρατός μέλος, με τη Φιλανδία προκειμένου για το πρώτο τομέα, ενώ για το σημείο 7 με τη Σουηδία, που είναι η έρευνα και η καινοτομία του 7. 80 είναι οι εμβληματικέ πρωτοβουλίες, τα προγράμματα στη Βαλτική που εφαρμόζονται. Τα έργα δηλαδή. Ορισμένα από αυτά ήδη βρίσκονται στο τελικό στάδιο και προετοιμάζουμε μια ευρύτατη θεώρηση του λεγόμενου προγράμματος δράσης που περιλαμβάνει όλα αυτά τα έργα Μετά από δύο έτη εφαρμογή, όπω σα είπα, η απόφαση του Συμβουλίου ήταν να γίνει η πρώτη αναθεώρηση. Ε, Και στην ουσία, βάση για την αναθεώρηση ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στις 22 Ιουνίου κατέθεσε μια ευρύτατη έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βαλτική. Και αυτή ήταν η βάση για την Πολωνική Προεδρία για να αρχίσει να προετοιμάζει την αναθεώρηση στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα στοιχεία για να σας πω πώς προετοιμάσαμε την ε, αναθεώρηση. Ποια ήταν τα βασικά ε, δεδομένα που εντόπισε, τα βασικά ευρήματα θέλετε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνούσαν πάρα πολύ με τα όσα εμείς ε, διαπιστώσαμε ως Προεδρία. Ε, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που ε, καθημερινά αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα της Βαλτικής, ότι βρέχονται από τη Βαλτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τι ε, διαπιστώνει και περιγράφει ως βασικά επιτεύγματα. Πρώτον, νέα έργα. Ή δίνεται μια νέα πνοή στα υφιστάμενα. Όπως γνωρίζετε η δινεται μια νεα απνοη θάλασσα, ακόμα και πριν τη στρατηγική, ήταν ε, πάρα πολύ καλή στη διεθνή συνεργασία και διεθνή και περιφερειακή και εθνική φορείς ασχολούνται με τη συνεργασία των χωρών της Βαλτικής. Υπήρχε μια πιο εργασία, ένα πλαίσιο δεδομένο και ακόμα και δύο χρόνια αργότερα βλέπουμε ότι το δυναμικό της περιοχής μας ε, και της περιφέρειας γενικότερα δεν έχει, πώς να το πω, εξαντληθεί η στρατηγική βοήθησε, τόνωσε, ενίσχυσε τη συνεργασία. Δημιούργησε νέα δίκτυα για ε, περισσότερη συνοχή και καλύτερη ανάπτυξη πολιτικής. Επίσης, ε, ενισχύθηκε η συνεργασία και με άλλα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευθυγραμμίστηκε κάπως η χρηματοδότηση με άλλες χρηματοδοτικές ε, πρωτοβουλίες. Συνεργαζόμαστε και με τη Ρωσία και με το CBSS ή το Βόρειο Σύμφωνο Υπουργών και ε, άλλους τοπικούς φορείς. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά νέα έργα Επιτρέψτε μου να σας τα παρουσιάσω, όχι σε λεπτομέρειες βεβαίως, απλώς για να σας δείξω ε, τι ε, έχει προκύψει. Για παράδειγμα, ε, προγράμματα για τους αγρότες που λέγεται Baltic Deal ή σχέδια για την καθαρή ναυσιπλοεία για να μειώνεται η ρήπανση από τα σκάφη. Επίσης, Balta DAP, μια μελέτη σκοπιμότητας για το LNG. Γενικά βλέπετε διάφορα προγράμματα που τονώνουν την καινοτομία, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα κλάστερ στη συνεργασία για την έρευνα. Ε, πολύ σημαντικό είναι το Scan Balt Health Port για την υγεία ή ένα άλλο πρόγραμμα για τις μεταφορές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και κάποιες συστάσεις που βλέπετε σε αυτή εδώ τη διαφάνεια. Πρώτον, για να πετύχει η στρατηγική για τη βαλτική θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί αυτή η ε, ε, πνοή που έχει δοθεί στο πρόγραμμα, αυτή η δυναμική και η στρατηγική και η πολιτική υποστήριξη. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί σε λίγο θα σας πω, εμείς τη έχουμε διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της αναθεώρησής μας. Είναι πάρα πολύ Ε, κοινή η εκτίμηση των ενδιαφερομένων για τα ζητήματα και τα προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη δέσμευση, στόχοι ε, και μέθοδοι ε, χειροπιαστές για την αποτίμηση του προγράμματος. Αυτό πραγματικά ήταν από τα σημαντικότερα διδάγματα της τελευταίας διετίας. Όταν δημιουργήθηκε η στρατηγική αυτή, δεν είχε ένα σύστημα στόχων και δικτών για να μπορεί κανείς να μετράει την εφαρμογή της. Και τώρα προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό και να ορίσουμε ένα κατάλογο στόχων ε, στην ομάδα εργασίας μας ε, για να υπάρχει μια καταμέτρηση. Επίσης υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας και εσωτερικής και εξωτερικής. Και θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό αφορά και το ευρύ αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των φορέων, των κρατών μελών, των ε, θεσμικών οργάνων, αλλά και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ τους, στο εσωτερικό της. Επίσης, υπάρχει και ένα ζήτημα προφανώς χρηματοδότησης. Θα πρέπει ε, να συγκεράσουμε τη χρηματοδότηση με την τεχνική υποστήριξη και βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα για τους συντονιστές των ε, τομέων προτεραιοτήτων. Now, a few sentences about the review process as such. Uh, when Poland was preparing for... Για την αναθεώρηση αυτή καθ' αυτή, η Πολωνία όταν προετοιμαζόταν να αναλάβει την Προεδρία uh, uh, είχε σκεφτεί πώς θα κάνει αυτή την αναθεώρηση. Έγιναν πολλές πολιτικές διαβουλεύσεις με ε, πολλούς φορείς και παράγοντες από νωρίς. Τον Απρίλιο άρχισαν οι πρώτες διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο και με ε, υπευθύνου διαφόρων έργων, διαφόρων προγραμμάτων σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων. Στην Πολωνία αυτό είναι ζήτημα που αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών. αλλά δεν ε, είχαμε ε, πρώτερη εμπειρία ε, πρακτικής εφαρμογής υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων. Λοιπόν, μετά τις διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο είχαμε σειρά διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη και της περιοχής βεβαίως της Βαλτικής, αλλά και εκτός με την Νορβηγία και την Ισλανδία και άλλους τέρους που είναι σημαντικοί για την περιφέρεια αυτή. Επίσης, Προσπαθήσαμε να έχουμε, να διαβουλεύσει και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα τη χαρά να συναντηθώ με ε, ε, τη διακομματική ομάδα, το Intergroup δηλαδή του Κοινοβουλίου για τη Βαλτική. Επίσης προσπαθήσαμε να ε, συλλέξουμε και τις γνώμες και τις γνωμοδοτήσεις της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής και συνεργασίας της Επιτροπής Περιφερειών. Βλέπετε ε, στη διαφάνεια τις διαβουλεύσεις αυτές. Ποια ήταν τα κύρια ευρήματα τώρα στις δύο επόμενες διαφάνειες. Θα διαπιστώσετε ότι πάρα πολλοί συμφωνούν με τα όσα διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, the report of, uh, Και αυτά που αναφέρει στην έκθεσή της της 22 Ιουνίου Τα βασικά θέματα που έχουν εντοπίσει και επισημάνει οι ε, ενδιαφερόμενοι και ενεχόμενοι για βελτιώσεις, πρώτα απ' όλα είναι η πολιτική υποστήριξη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα και το τονίζω. Δεν αρκεί η πολιτική υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει και σε επίπεδο περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να υπάρχει υποστήριξη. Ε, επίσης, ε, ο ρόλος του καθενός θα πρέπει να διευκρινιστεί και να ενισχυθεί έτσι και αλλιώς είναι περίπλοκη αυτή η στρατηγική στην οργάνωσή της, οπότε θα πρέπει να ε, ορίζεται καλύτερα ο ρόλος του καθενός, ε, των προτεραιοτήτων, των τομέων, των συντονιστών. Ένα άλλο θέμα είναι το σύστημα ακριβώς ε, αξιολόγησης που να βασίζεται σε στόχους και σε δείκτες μετρήσιμους. Επίσης καλύτερη χρηματοδότηση ή καλύτερο συντονισμό στη χρηματοδότηση. Γιατί αυτή τη στιγμή που προετοιμάζουμε το επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις μακροοικονομικές στρατηγικές. Είναι η πρώτη φορά που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μακροχρόνιο σχεδιασμό και θα πρέπει ε, να γίνει σωστά η προετοιμασία. Επίσης, βελτίωση της επικοινωνίας και της προβολής, συμμετοχή διαφόρων τομεακών πολιτικών και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Όπως γνωρίζετε, μετά από τα δύο πρώτα χρόνια διαπιστώσαμε ότι η στρατηγική αυτή βασίζεται και εντάσσεται κυρίως στην πολιτική συνοχή. Εμείς θέλουμε να το διευρύνουμε αυτό, να συμμετέχουν και άλλοι τομείς. Παράδειγμα, υποδομές, μεταφορές, ενέργεια, καινοτομία, έρευνα κτλ. Άλλο θέμα. Οι συνέργειες, η συνεργασία δηλαδή μεταξύ διαφόρων ε, φορέων της στρατηγικής αυτής και άλλες πλατφόρμες συνεργασίας στη Βαλτική. Όπως γνωρίζετε, στην περιφέρεια της Βαλτικής υπάρχουν διάφορα φόρα, το CSS, το ε, Βόρειο Συμβούλιο, το HealthCo. Είναι πολλά τα προγράμματα και θέλουμε καλύτερα να συντονίζονται, να συνδυάζονται. Υπάρχουν δίκτυα, δεν είναι νέες δομές και θα πρέπει καλύτερα να συνεργαζόμαστε, να συντονιζόμαστε ε, για να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα χωρίς επικαλύψεις. Επίσης, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Γνωρίζετε ότι αυτό τον καιρό έχουμε δύο στρατηγικές, η για το, τη Βαλτική θάλασσα, αλλά και έχουμε και για το Δούναβι. και θα πρέπει να επιζητήσουμε τη συνεργασία. Ακόμα και σε επίπεδο ανταλλαγή εμπειριών, ε, συνεργασία, δημιουργία δικτύων κτλ. The review, Όπως σας είπα, στην αρχή η αναθεώρηση βασίζεται στη συνεργασία στο ιστορικό του Συμβουλίου θεσπίσαμε ξανά μια ομάδα που λέγεται Friends of Presidents, οι φίλοι της Προεδρίας, ε, που προετοιμάζει τα συμπεράσματα για τη βελτίωση της στρατηγικής. Ε, συστήθηκε η ομάδα αυτή τον Ιούλιο και θα εργαστεί μέχρι αρχές Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα πάμε στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων στο ΚΟΡΕΠΕΡ για να εγκριθούν τα συμπεράσματα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, ως Προεδρία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέτος το BDF, το δεύτερο ετήσιο φόρουμ για τη Βαλτική, θα φιλοξενηθεί στο Γκτάνσκ, όπου συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την περιφέρεια και το Δήμο του Γκτάνσκ. 24 με 26 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα αυτή η πρωτοβουλία και θα ήθελα επευκαιρία να σας καλέσω. Uh, ε, θέλουμε εκεί να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι όσοι ασχολούνται με τη στρατηγική αυτή στην καθημερινή τους ε, εργασία και αυτό το φόρουμ θα είναι ένας χώρος συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων που θα καταλήξει σε πάρα πολύ πρακτικά συμπεράσματα ε, και συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση αυτής της στρατηγικής. Και ελπίζουμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τελικά να έχουμε μια σειρά πρακτικών συστάσεων και προτάσεων για μια αναθεωρημένη επικοινωνία και ανακοίνωση μάλλον για τη στρατηγική αυτή που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 όπως ελπίζουμε υπό δανική προεδρία. Άλλη μια χώρα της Βαλτικής που προεδρεύει για να ολοκληρώσει ε, το έργο μας. Σταματώ εδώ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με χαρά να απαντήσω αν έχετε κάποιες ερώτηση. Ευχαριστώ. Uh, very much for this σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τόσο ολοκληρωμένη ε, εισήγηση για αυτά τα τόσο στρατηγική σημασία θέματα. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον κύριο Μπελάρντι να μιλήσει για την ε, μακροπεριφέρεια ε, Αδριατική Ιωνίου και μετά θα έχουμε τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητάς. Παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και μεταφέρω και τον χαιρετισμό του Προέδρου της ε, Περιφέρειας, ο οποίος δυστυχώς ε, δεν μπορεί να είναι εδώ, βρίσκεται στην Ρώμη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο Φρανσουά Αλφονσί, καθώς επίσης και την πρόεδρο Χιούμπνερ, οι, οποία, οποίοι μας κάλεσαν εδώ για να μιλήσουμε για αυτή την μακροπεριφέρεια.

στην ε, Βαλτική προϋπήρχε ένα δίκτυο ε, σχέσεων αλλά και στην ε, Αδριατική κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας βάσει των οποίων προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας βεβαίως το πλαίσιο το ευρωπαϊκό και λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες με στόχο την ενίσχυση της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται εδώ και αιώνε από κοινού πολιτιστικού και οικονομικούς δεσμού και πρόσφατα από μεγάλε προσπάθειε εν ολοκλήρωσης όπως ας πούμε αυτή τη Αδριατικής Ιωνίου ε, μέσα από συνεργασία των εμπορικών επιμελητηρίων κλπ. Πέρα από πολλά δίκτυα τα οποία αφορούν πολιτιστικά θέματα έχουν λοιπόν δημιουργηθεί ε, και άλλοι δεσμοί πολιτιστικά αναφέραμε βεβαίως σε κάθε μορφή πολιτισμού. Η πρωτοβουλία γεννήθηκε, δημιουργήθηκε το 2000 στην Αγκώνα ε, ε, και είχε κύριο στόχο την συνεργασία για την ασφάλεια της Αδριατικής και της Ιωνίου. Ε, και ε, μεταξύ, εκτός της Ελλάδας και της Ιταλίας ε, υπάρχουν, συνεργάζονται επίσης και όλες οι άλλες όμορες περιοχές, πρόσφατα δε και το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Υπάρχει η μόνιμη γραμματεία του, της Αγκώνα που και μέχρι το 2012 η Προεδρία ανήκει στη Σερβία. Ο στόχος ε, της πρωτοβουλίας για την οποία γίνεται λόγος ε, είναι να βελτιώσει τη συνεργασία στην ε, Μεσόγειο, σε αυτή την περιοχή της Μεσογείου, μέσα από συνεργασία όσον αφορά το περιβάλλον, τις θαλάσσιες μεταφορές, τα πανεπιστήμια και άλλα. Θεωρούμε ότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν πυλώνες ισχυρούς για την ανάπτυξη μιας μακροπεριφερειακής πολιτικής για την Αδριατική και το Ιόνιο, στα πλαίσια του οποίου η μακροπεριφέρεια θέλει να προωθήσει την εταιρική σχέση μεταξύ των μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι στα πλαίσια της ε, μακροπεριφέρειας το 2010 τα 8 κράτη-μέλη προσυπέγραψαν τρία πρωτόκολλα συνεργασίας ε, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, τον τουρισμό και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Την 5η Μαΐου του 2010 στην Αγκώνα και 13 Μαΐου του 2011 οι ε, ε, Υπουργοί Εξωτερικών των 8 χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία προσυπέγραψαν δύο δηλώσεις ε, βάσει των οποίων δεσμεύονται ρητά να αναγνωρίσουν την μακροπεριφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, το, για την Αδριατική και το Ιόνιο. Το δεύτερο φόρουμ είναι αυτό των πόλεων ε, της Αδριατικής και, ε, ε, του Ιωνίου. Στη δημιουργήθηκε το 1995 και συμμετέχουν πάνω από 350 πόλεις της περιοχής. Στόχος είναι να αναπτύξουν τη συνεργασία όσον αφορά πολιτιστική, οικονομική, εμπορική συνεργασία. Υπάρχει επίσης το Φόρουμ των Επιμελητηρίων που δημιουργήθηκε το 2001 και έχει 36 μέλη. η ε, περιφέρεια την οποία καλύπτουν αυτά τα εμπορικά επιμελητήρια αποτελεί ε, ένα πάρα πολύ μεγάλο πουλ επιχειρήσεων, πάνω από ένα εκατομμύριο ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με μεγάλο τζίρο καθώς επίσης και με μεγάλη γεωγραφική έκταση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικό στοιχείο για την, για την συνοχή της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης συνεργασία ε, μεταξύ των πανεπιστημίων και προσφάτως έγινε μέλος και η Μακεδονία, λέει ο μιλητής. Ε, δημιουργήθηκε ε, προσφάτως αυτή η ιδέα έτσι ώστε να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ των πανεπιστημίων και να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ε, επίσης πρόσφατα δημιουργήθηκε και άλλο ένα ε, δίκτυο το οποίο αφορά τις έξι χώρες που βρέχονται από την ε, Μεσόγειο. Δημιουργήθηκε τον προηγούμενο χρόνο έτσι ώστε να βελτιώσει την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βελτιώσει επίσης την αμοιβαία κατανόηση των κατοικούντων στις περιοχές αυτές. Όσον αφορά την διακυβέρνηση, αναφέρεται ρητά στι συνθήκε Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν είναι δυνατόν ε, να ε, υπάρξει εφαρμογή της διακυβέρνησης στο επιθυμητό επίπεδο, εάν σε επίπεδο ε, περιφερειών δεν υπάρχει επίσης σωστή διακυβέρνηση. Κατά αυτήν την έννοια, η στρατηγική των μακροπεριφερειών αποτελεί καινοτόμα αντιμετώπιση τη περιφερειακή διακυβέρνηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί αηφόρο και ισορροπημένη ανάπτυξη ανάπτυξη καθίσταται δε σαφές ότι πρόκειται για λειτουργικές μακροπεριφέρειες, ε, δηλαδή συγκεκριμένες ε, εδαφικές ενότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινές, ε, που αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Τα διακυβέρματα δεν είναι κοινά και επομένως είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν κατά μόνας. Είναι πολύ πιο εύκολο από κοινού να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις οι οποίες κάθε μέρα γίνονται και περισσότερες. Βασιζόμαστε βεβαίως στη συνθήκη της Λισαβόνας και προσπαθούμε να διευκολύνουμε την είσοδο τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ε, μακροπεριφέρεια ε, της Αδριατικής και του Ιωνίου, ε, είναι μια λειτουργική περιφέρεια η οποία, η οποία συνδυάζει τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς που σκύβουν πάνω από κοινέ προβληματικές και που καταφέρνει να συνδυάσει χώρες οι οποίες είναι μέλη και χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θεσμικά ε, πρέπει να υπάρχει μια ε, συγκεκριμένη δομή, όμως οι κοινέ ε, δράσεις ε, ε, που έχουν οπωσδήποτε μία θεσμική βάση είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να βασιστούν σε υφιστάμενα προγράμματα. Γι' αυτό ακριβώς η περιφέρεια Αδριατικής Ιωνίου ασχολείται με συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα θέματα τα οποία κυρίως είναι προσφυλή στι στις χώρες μέλη. Και Βεβαίω, ασχολείται και με θέματα τα οποία απασχολούν τις χώρες και, ε, που βρίσκονται και προς Ανατολάς και προς δυσμάσα της περιφέρειας αυτής. Η μακροπεριφέρεια ε, έχει στόχο να διασυνδέσει καλύτερα τα εδάφη που την αποτελούν ε, και να προστατέψει βεβαίως το περιβάλλον κυρίως ε, τόσο στην ξηρά όσο και τα ιδιαίτερα ευάλωτα θαλάσσια περιβάλλοντα η Ιταλία με, την, με τις περιφέρειες Αδριατικής Ιωνίου, η Σλοβενία και η Ελλάδα καθώς επίσης και η Κροατία ε, που θα γίνει μέλος ε, σε τρία χρόνια, καθώς επίσης και η Βοσνία Ζεγοβίνη και άλλες δύο χώρες οι οποίες είναι ε, υποψήφιες, έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, 400.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ακτών. Πρόκειται λοιπόν για μια περιφέρεια η οποία ξεπερνάει την λεκάνη τη θαλάσσια λεκάνη και αποτελεί μια δυνατότητα δυνατότητα διασύνδεσης, ένα κρίκο διασύνδεσης ανάμεσα στους πολιτισμούς και τους πληθυσμούς που κατοικούν την ε, περιφέρεια αυτή. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια ανταλλαγών, απόψεων, πολιτιστικών συνηθιών, ε, εμπορίου, αγαθών, προϊόντων κτλ. Η προστασία των θαλασσίων υδάτων, κυρίως δε ε, των ακτών, οδηγεί σε μια πιο μεσογειακή προοπτική. Ε, και μπορεί να βοηθήσει στην σταθεροποίηση της ε, περιοχής. Υπενθυμίζω ότι ε, υπάρχουν, στην περιοχή υπάρχουν πολλές χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την ενέργεια και κτλ. Ε, αλλά ε, υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά εθνικά προγράμματα στους στόχους 1 και 2, περιφερειακά προγράμματα, καθώς επίσης και προγράμματα διασυνεργειακής συνεργασίας, ας πούμε, μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας κτλ. Πέρα από τις διεθνικές συνεργασίες υπάρχουν και άλλα ιδιαίτερα προγράμματα προγράμματα, ε, προγράμματα για τις αλπικές περιοχές, προγράμματα για την Μεσόγειο κτλ. Αντιθέτως, ε, τα TENS ε, φαίνεται ότι έχουν ξεχάσει την περιφέρεια αυτή πέρα από, τον, πέρα από τη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την Ελλάδα με την Ανατολική Ευρώπη. Η ιδέα της ύπαρξης της μακροπεριφέρειας Αντριατικής Ιωνίου ε, βασίζεται στα ωφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων, ε, τα ε, εθνικά κεφάλαια και τα ιδιωτικά κεφάλαια συνεργάζονται έτσι ώστε να υπάρξει μια ευρύτερη λογική, δηλαδή να μην υπάρχει μια περιοριστική και συσταλτική λογική διακυβερνητικών συνεργασιών από την αρχή του 2010 και σε στενή συνεργασία με το ε, Υπουργείο Εξωτερικών ε, της Ιταλίας καθώς επίσης και την πρωτοβουλία ε, της μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου η περιφέρεια της, των Μαρκών έχει ξεκινήσει μια ιδιαίτερη διαδικασία. Τον Μάρτιο του 2011 η Επιτροπή Περιφερειών δια της Αρμοδίας Επιτροπής της ε, έδωσε στην, ε, ανέθεσε μάλλον στην Περιφέρεια ε, Μάρκε την μελέτη, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με γνωμοδότηση όσον αφορά τη λειτουργία της μακροπεριφέρειας η πρώτη, ε, ε, η πρώτη ημερομηνία ήταν 4η Ιουλίου και ε, έγινε η πρώτη υποβολή, η πρώτη παρουσίαση μάλλον της έκθεσης και αργότερα θα υπάρξει η συζήτηση στην Ολομέλεια το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Ιουνίου 2011 στα συμπεράσματά του κάλεσε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν ε, την εργασία σε συνεργασία με την Επιτροπή για τη δημιουργία μελλοντικών μακροπεριφερειών ε, με συγκεκριμένη αναφορά στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Ε, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε επίσης να συντάξει γνωμοδότηση Τη πρωτοβουλίας μέχρι το τέλος 2011 για την ίδια μακροπεριφέρεια. Ταυτόχρονα ε, ενεργοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των ε, τοπικών περιφερειών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσα από πολλά συνέδρια, επαφές, συναντήσεις στα ε, κράτη-μέλη της ε, πρωτοβουλίας ε, από τις Ιταλικές περιφέρειες και από διάφορα φόρουμ τα οποία ενδιαφέρουν τις περιφέρειες. Στην ανακοίνωση που, στην οποία αναφέρθηκε και προηγουμένως και που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικού, Εξωτερικών αναφέρεται το ίδιο η σημασία ύπαρξης της μακροπεριφέρειας. Τα στις 23 Ιουνίου του 2011 στην, ε, στο φόρουμ των αυτόνομων περιφερειών της Ιταλίας ε, στα συμπεράσματα αναφέρεται ρητά η δέσμευση στήριξης ε, της μακροπεριφέρειας και επίσης η έκθεση η οποία οργανώθηκε στην Αγκώνα τέλη Αυγούστου και στην οποία, στην οποία ήταν παρούσες όλες οι χώρες της μακροπεριφέρειας η, τα, τα εργαστήρια, τα workshops τα οποία πολύ σύντομα θα οργανωθούν συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ιταλίας, της Σερβίας και άλλων όμορων ε, κρατών που έχει οργανωθεί την 25η Οκτωβρίου στην Αγκώνα, καθώς επίσης και άλλα σεμινάρια τα οποία προβλέπονται ε, για τον Δεκέμβριο μαρτυρούν ε, την μεγάλη ευαισθητοποίηση ε, των χωρών όσον αφορά την μακροπεριφέρεια. Ε, ε, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει συγκεκριμένη θεσμοθετημένη εντολή στην Κομισιόν όσον αφορά αυτή την μακροπεριφέρεια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνοχή και σε οικονομικό και σε πολιτισ... θεσμικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, μακροπεριφέρεια Αδριατικής και ε, Ιωνίου μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο όχι μονάχα για τις ενδιαφερόμενες περιοχές αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να οδηγήσει σε αηφόρο ανάπτυξη και τέλος να οδηγήσει οδηγήσει στην κάλυψη των προϋποθέσεων της Ατζέντα Ευρώπη 2020. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη ανοίγεται πλέον προς τα, δυτικά, προς τα ανατολικά, ε, ε, δυτικά, προς τα δυτικά Βαλκάνια. Και κατά αυτή την έννοια ε, οι περιφέρειες αυτές οι οποίες έχουν, βρίσκονται πλέον σε προενταξιακές διαδικασίες και οι οποίες αποτελούν μέλος μέρος της μακροπεριφέρειας μπορούν να βοηθηθούν στη διαδικασία εκδημοκρατίας τους και στη διαδικασία γυτνίασης ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ε, βάσει των δραστηριοτήτων και των δράσεων της μακροπεριφέρειας να στηρίξουμε την ανάπτυξη, την αηφόρο ανάπτυξη. Θέλουμε ε, η στρατηγική για την μακροπεριφέρεια να είναι ε, συγκεκριμένη, να έχει έμπνευση για το μέλλον έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη μέγιστη δυνατή ολοκλήρωση πολιτιστική, οικονομική, εμπορική κλπ. Όπως έλεγε προηγουμένως η συνάδελφος ε, για την Βαλτική και τον Δούναβη, αλλά και η δική μας στρατηγική για την δική μας μακροπεριφέρεια μπορούν ε, να οδηγήσουν και σε δημιουργία σημαντικών υποδομών, έτσι όπως ε, αναφέρεται στο σημείο 18 της ανακοίνωσης του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2011 και μπορούν να αποτελέσουν στην συνεργασία τους έναν ιδεώδη άξονα ε, βορρά-νότου. Η πρόσβαση προς την νότιο-ανατολική Ευρώπη ξεκινώντας από το βορρά ε, με τη δημιουργία τέτοιων υποδομών θα διευκολύνεται σημαντικά οι εταίροι θα ε, ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, τις οποίες θα επιλέξουν αν και ήδη ξέρουμε ότι οι επικοινωνίες, ε, οι θαλάσσιοι λεωφόροι, η ασφαλής ναυσιπλοεία είναι, αποτελούν ήδη πρώτες προτεραιότητες. Για, όλα, για όλους αυτούς τους λόγους που ήδη ανέφερα θεωρούμε ότι ε, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ε, δε η πολιτική συνοχή για την περίοδο μετά το 2013 θα πρέπει οπωσδήποτε να εντάξει ε, τις μακροπεριφ... τους μακροπεριφερειακούς στόχους και τις μακροπεριφερειακές συνεργασίες κυρίως αναφερόμενοι στις διασυνοριακές συνεργασίες. Και για την προγραμματική περίοδο 14-20 θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να διευκολυνθούν αυτές οι στρατηγικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει και των δηλώσεων και των βουλήσεων που ε, ε, ήδη έχουν εκφραστεί από τις χώρες μέλη και λαμβάνοντας υπόψη και την στρατηγική αξία της ολοκλήρωσης της ενταξιακής πορείας διαφόρων χωρών καθώς επίσης και της ανάγκης υλοποίησης και ολοκληρωμένης ναυτικής και θαλάσσιας πολιτικής και πολιτικής μεταφορών. Είναι αναγκαίο λέω να ε, εφαρμόσει ολοκληρωμένες πολιτικές και για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Κατά την ίδια έννοια θα ήθελα να σας υποβάλω ε, το ενδεχόμενο στις Βρυξέλλες να γίνει ε, η ετήσια συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου που προβλέπεται για τον Απρίλιο-Μάιο του 2012. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπελάρτη. Συζήτηση. Κύριος Αλφονσί, εισηγητής της εκθέσης πρωτοβουλίας και στη συνέχεια δεξιόνις κοιόδης θέλουν τον λόγο. Κύριος Αλφονσή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ καταρχήν τους προλαλήσαντες για τη σαφήνεια και τα συγκεκριμένα μηνύματα από την εμπειρία καταρχήν της Βαλτικής γιατί μετά από δύο χρόνια μόνο έχουμε ήδη απτά αποτελέσματα. Έχουμε μία μέθοδο εργασίας και συγκεκριμένη απτή υπεραξία χάρη στην μακρο στρατηγική. Τη στρατηγική ήταν μακροπεριφέρεια. Η διαδικασία αυτή της Βαλτικής και ο ενθουσιασμός δείχνουν πόσο προχωράει η ευρωπαϊκή ιδέα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας. Ως προς την Μεσόγειο και εκεί υπάρχει ελπίδα, υπάρχει κινητοποίηση. Σήμερα στο επίπεδο των μακροπεριφερειών που έχουν στόχο την εδαφική ανάπτυξη, βλέπουμε μια προσδοκία βάσιμη. Από εδώ και πέρα, στο πλαίσιο των στόχων του 2020, αυτά ας ληφθούν υπόψη, διότι πρόκειται για προσδοκίες και κινητοποίηση στις περιφερειές μας που πρέπει να ληφθούν υπόψη ακριβώς από την ευρωπαϊκή πολιτική για μας με βάση τις πρώτες εμπειρίες ήρθε η ώρα να καθορίσουμε το μέλλον της στρατηγικής μας για τις μακροπεριφέρειες. Πρέπει να καταστρώσουμε λοιπόν μια ειδική στρατηγική. Διότι από εδώ και πέρα Έχουμε μια Σουηδική Προεδρία, μια Πολωνική Προεδρία. Το θέμα είναι, πέραν αυτών, ποια θα είναι η κινητήρια δύναμη η οποία θα υλοποιήσει αυτές, αυτή την στρατηγική. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις μακροπεριφέρειες στην γενικότερη στρατηγική μας. Αυτό πρέπει να είναι και το αντικείμενο του διαλόγου, εξού και η έκθεση πρωτοβουλία που θα παρουσιάσω τον επόμενο μήνα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε περίπου πού πηγαίνουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά τους περιορισμούς της σημερινής πολιτικής και να δούμε από εκεί πέρα τι χρειάζεται να κάνουμε. Η στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα γενικότερο ακόμη πλαίσιο, είναι προϊόν μάλλον αυτοσχεδιασμού η Επιτροπή των Περιφερειών, η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο έκαναν ό,τι μπορούσαν με καλή θέληση και ενθουσιασμό αλλά χωρίς να διαθέσουν τους πόρους που απαιτεί η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, τώρα ακριβώ που συζητούμε την περίοδο 14-20, να προσπαθήσουμε να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις με τρόπο επιπλέον για να καταστρώσουμε και μια καλύτερη στρατηγική για την Ευρώπη γενικότερα. Εγώ θα πω δύο λόγια για την ε, Μεσόγειο. Μεταξύ άλλων, διότι πλήττεται περισσότερο από την κρίση. Πρέπει λέει, λοιπόν προς τη Μεσόγειο να στείλουμε μήνυματα αισιοδοξία Έχουμε την κρίση στην Ελλάδα, προς την οποία πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Η αλληλεγγύη αυτή είναι παρούσα, αλλά πρέπει να στείλουμε και μηνύματα που έχουν σχέση με την αυστηρή εκτέλεση του προπολογισμού. Γιατί πρέπει να είμαστε αυστηροί έναντι των κυβερνήσεων των χωρών μελών. Γενικότερα. Τώρα, αν θέλουμε η ιδέα της Ευρώπης να λάβει μια επιπλέον όθηση, το μήνυμα πρέπει να είναι θετικό, επικοδομητικό. Και εδώ έχουμε την ευκαιρία, στο πλαίσιο δηλαδή, τη πολιτικής για τη Μεσόγειο, να στείλουμε ένα αισιοδόξο μήνυμα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μόνο η βόρεια ακτή τη Μεσογείου. Το χρειάζεται και η νότια ακτή, στην οποία συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα τελευταία. Σε αυτέ λοιπόν τι προσδοκίε και στις προσδοκίε της νότιας ακτής της Μεσογείου πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση για περισσότερη ανάπτυξη σε όλη τη Μεσόγειο και στο Βορρά και στο Νότο. Εν κατακλείδη, η Μεσόγειος είναι ένας ενιαίος χώρος. Χαρακτηρίζεται από ένα κοινό σημείο, το γνωστό μεσογειακό κλίμα. Όλοι ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Βλέπετε, αντίστοιχα, αν όχι ίδια αγροτικά προϊόντα, ίδια περιβαλλοντικά προβλήματα, πυρκαγιές για παράδειγμα στα δάση. Για να μην μιλήσουμε και για τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Ο πολιτισμός και η ζωή γεννήθηκαν στη Μεσόγειο. Κατά τα άλλα, μιλάμε για μια μεγάλη περιοχή με μεγάλες αποστάσεις από την Ανατολή ε, στη Δύση. Τώρα μιλούμε βεβαίως εδώ για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου που χαρακτηρίζεται από τη δική της προβληματική. Θα πω λοιπόν ξανά ότι αυτές οι στρατηγικές αφορούν βεβαίως τη βάση αλλά έχουν και μια γενικότερη ευρύτερη διάσταση. Εδώ ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δρομολογήσει το σχετικό διάλογο, το λεφτό και προς την Κομισιόν, γιατί αν η στρατηγική για την μακροπεριφέρεια ενταχθεί στη γενικότερη πολιτική μας, τότε θα είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε το έργο αυτό στο χρόνο, να θεσπίσουμε τις προτεραιότητές μας και ο διάλογος να γίνει πιο δομημένος ακριβώς επειδή εμπλέκονται πολλοί εταίροι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν από τώρα να πούμε ακριβώς τι θέλουμε και όταν έρθει η ώρα να μπορέσουμε να κινηθούμε με βάση συγκεκριμένε προτεραιότητες. Να εξετάσουμε επίση το θέμα της διακυβέρνησης, γιατί κανένα έργο δεν προχωρά χωρίς σωστή διακυβέρνηση. Είμαστε στη φάση λοιπόν την προκαταρκτική. Καλό όλους να δείξουμε μεγαλύτερο ενθουσιασμό και περισσότερη οργάνωση. Ευχαριστώ πολύ. Χιούμπνερ. Ευχαριστώ. Τόμας Ντόιτς, ο πρώτος σκιώδης. Παρακαλώ. előadást. Természetesen szeretném Ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές, τους ομιλητές ε, για τα όσα μας είπαν. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε και θα βοηθήσει και τον εισηγητή και σε λίγο καιρό θα έχουμε και το έγγραφο εργασία. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια ε, σχετικά με τη σημερινή μας συζήτηση. Η Πολωνική Προεδρία μίλησε για τη στρατηγική της Βαλτικής. Και ξεκαθάρισε ότι η έκθεση αυτή ε, συζητείται και στο Συμβούλιο και θέλουν, λέει, να συνδυάσουν τη στρατηγική της Βαλτικής με τη στρατηγική του Δούναβεως και το 2013 να γίνει μια αξιολόγηση βάσει κάποιων κριτήριων. Δεν θα ήταν καλό να έχει τη δυνατότητα έτσι και το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας και το Συμβούλιο να βασίζονται σε κάποια κριτήρια και μέχρι το 2013 να μπορούν να συγκρίνουν, να εκτιμήσουν, να αναθεωρήσουν, να αξιολογήσουν αυτές τις δύο στρατηγικές. Η έκθεση του συναδέλφου Αλφόνση ελπίζω να μας επιτρέψει να σκεφτούμε για το μέλλον των μακροπεριφερειών να είναι όμως ενιαία συστήματα αρχών και κριτηρίων και να έχουμε ένα μπούσουλα για να μπορούμε να πορευόμαστε. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. παρατήρηση δεύτερη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί η πρωτοβουλία για τη στρατηγική του Δουνάβεως και της Βαλτικής μπορεί να ήταν επιτυχής, αλλά ε, χρειάζεται μια συγκράτηση εδώ τώρα, να μην ε, μπούμε σε μια μόδα ε, και δημιουργήσουμε νέα ε, χιονοστιβάδα, συνέχεια όλο και περισσότερες μακροπεριφέρεια και στρατηγικές. Στο παρελθόν Υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά ορισμένες ήταν ε, επειδή είχαν γίνει του σειρμού οι πολιτικές και οι στρατηγικές και πολλαπλασιάστηκαν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι δύο μακροπεριφερειακές στρατηγικές να ε, ειδωθούν ως ένα ενιαίο σύνολο με συγκεκριμένα κριτήρια, αρχές ε, για την αξιολόγηση. Και ένα τρίτο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ πολύ σημαντικό Στη νέα φάση της πολιτικής συνοχής και στη νέα προγραμματική φάση θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες αρχές για την εκπόνηση τέτοιων πολιτικών στο μέλλον. Θα ήθελα να αποφύγω δηλαδή μια κατάσταση όπου και επιτρέψτε μου τώρα ίσως να υπερβάλλω και λίγο. Θέλω, λέω, να αποφύγουμε μια κατάσταση τύπου Κροατίας. Υπήρχαν κάποιες αρχές, κάποιοι όροι για τις διαπραγματεύσεις, αλλά ε, τράβηξαν πολύ σε μάκρος αυτές οι διαπραγματεύσεις και τελικά οι αποφάσεις επολύφθηκαν ήταν ε, πολιτικές. Ο καθένας βλέπει λοιπόν ε, το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο και τελικά τα πολιτικά στοιχεία επικράτησαν απέναντι των τεχνικό Βεβαίω χρειάζεται πάντα μια πολιτική βούληση ε, όταν έρχεσαι να δικαιολογήσει μια στρατηγική, μια πολιτική. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κανόνες, σύστημα, κριτήρια, αρχές για να μην γεμίσουμε μακροπεριφερειακές στρατηγικές. να είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια και να, να είναι δικαιολογημένη η ε, δημιουργία νέα τέτοια περιφέρεια, όχι απλώ επειδή έγινε μόδα. Ευχαριστώ. Ο χρόνο πιέζει. Παρακαλώ, Σκιώδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές ε, που καταδεικνύουν μέσω των εισηγήσεων τους ότι ε, μπορεί το εργαλείο αυτό των μακροπεριφερειών να είναι ένα καλό εργαλείο επίτευξης διαφόρων στόχων μεταξύ των οποίων και ο στόχος που περισσότερο προσφυλής είναι για μας ε, στην Επιτροπή μας δηλαδή να γίνει όλο και πιο συνεκτική και όλο και πιο ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Κατά αυτή την έννοια πιστεύω ότι πολύ καλά έπραξε ο εισηγητής μας Φρανσουά Αλφονσί ε, που προσπάθησε να εξεύρει κάποιες αποφάσεις και υπό το φως των ε, στρατηγικών της περιφέρειας της Βαλτικής αφενός και αφετέρου μια σειρά ετοιμάτων που μου φαίνονται ήδη ε, καλά διαρθρωμένες όσον αφορά την, ε, ε, την επιθυμία να γίνουν ε, βήματα προς τα εμπρός σε συντονισμό και σε συνέργεια με την συνολική και συνεκτική πολιτική της Ευρώπης και στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά αυτή την έννοια θα πρέπει πρώτον να αποφύγουμε την επικάλυψη ε, ε, δομών και διαρθρώσεων. Γι' αυτό λοιπόν αυτά, αυτές οι μακροπεριφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ε, για τους, για τους πολίτες και να αποφύγουμε λοιπόν την δημιουργία νέων επικαλυπτόμενων διαρθρώσεων. Επίσης, Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη κρίση την οποία διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό ως Ευρώπη να δείξουμε ένα πρόσωπο το που δεν θα είναι μονάχα αυτό της διαρκώς ε, μεγαλύτερης απέτησης για μεγαλύτερη ε, λιτότητα. Ε, και επομένως να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και σε αυτά τα προβλήματα των πολιτών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει οι αποφάσεις που θα πάρουμε ε, θα πρέπει λέω να λαμβάνουν υπόψη τους ε, αυτά τα στοιχεία και αυτές τις προτάσεις και επομένως και ο Σέλφος Αλφονσί να λάβει υπόψη του αυτού του είδους τη διακυβέρνηση που θα παίρνει, θα υπολογίζει τις τοπικές στρατηγικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μιχαήλ δεν είναι εδώ. Άρα, Μαρή Τερέζη Σάντσες Σμιτ, σε πρώτη φάση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εντάχει, καταρχήν εκφράζω την ικανοποίησή μου για τον διάλογο αυτό, για τις μακροπεριφέρειες. Πολύ σημαντικός, εξαιρετικά εργαλεία για τον συντονισμό των προγραμμάτων σε ευρύτερη κλίμακα. Να επενθυμίσω τον διεθνικό χαρακτήρα του στόχου 3. Ο σχετικός διάλογος μπορεί να βοηθήσει και εδώ. Και θα ήθελα, όπως άλλωστε έπραξα και στην έκθεσή μου για την εδαφική συνεργασία, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιου πληθωρισμού τέτοιων στρατηγικών περιτών Ας επικεντρωθούμε λοιπόν ε, στην Μεσόγειο για παράδειγμα. η εξέλιξη στον αραβικό κόσμο το επιβάλλον Ο κ. Αλφόνση έστειλε ένα εξαιρετικά επικοδομητικό μήνυμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, συμφωνώ, να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα, προκειμένου. Μετά, στην Μεσόγειο, πρέπει να συνεργαστούμε με το πρόγραμμα MED, στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας. Και όσον αφορά τις προτεραιότητες, τις πρωτοβουλίες για την Μεσόγειο, πρόκειται για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εξαιρετικά χρήσιμες. Να τονίσω τέλος ένα ερώτημα, ένα ζήτημα το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό και το οποίο χρήζει προσοχής. Πώς θα παροτρύνουμε, θα παρακινήσουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να επενδύσουν ακριβώς σε αυτήν την στρατηγική της μακροπεριφέρειας. Κατσίφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Χαίρομαι που συζητούμε το θέμα. Είμαι υπέρ των μακροπεριφερειών και εγώ. Χαίρομαι που γίνονται πράγματα προς τα εμπρός, προς τη σωστή κατεύθυνση. Βρέθηκαν επικοδομητικές λύσεις χάρη στην επίσημη αλλά και άτυπη συνεργασία. Εν τέλει, έτσι ξεκίνησαν διάφορες συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα. Έχει σημασία από εδώ και πέρα να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα φέρνει πιο κοντά περιοχές που τους άλλους συνεργάζονταν εδώ και πολλά χρόνια. Με τον κύριο Ντόιτς όμως επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Είπε ότι πρέπει να περιορίσουμε τις δυνατότητες δημιουργίας επιπλέον μακροπεριφερειών. Μα γιατί? Ίσα ίσα. Τέτοιες συνεργασίες υπάρχουν εδώ και 10 χρόνια και περισσότερα. Γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες να μην ενσωματωθούν ακριβώς στο σύστημα αυτού των μακροπεριφερειών. Συμφωνώ από την άλλη πλευρά με τον εισηγητή ότι αυτό πρέπει να γίνει βάσει συγκεκριμένων όμως κριτηρίων. Ακούσαμε από την εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας σχόλια για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Σύμφωνοι. Το ερώτημα μου όμως είναι εάν στη διάρκεια της κρίσης έχουμε λόγο να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα για αυτές τις μακροπεριφέρειες. Το λέω αυτό διότι η εδαφική διάσταση είναι μια στρατηγική προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και οι μακροπεριφέρειες όμως το ίδιο για την περίοδο μετά το 2013. Αυτό τώρα τι σημαίνει. Σημειώστε πάντως αυτό να κρατήσουμε ότι υπάρχουν μακροπεριφέρειες που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ σύντομο. Κέλλη. Ενδιαφέρουσε παρουσιάσει. Γιατί ασχολούμαι με την στρατηγική για τον Ατλαντικό και ξέρω ότι όλα αυτά θα είναι υποφελή. Θα δημιουργήσουν δηλαδή προσθεμένη αξία. Όσον αφορά την Βαλτική, ακούσαμε για 15 προτεραιότητες, 8 εμβληματικά σχέδια και γνωρίζω λεπτομέρειε για μερικά από αυτά. Θα ήθελα να ακούσω όμω περισσότερα για να καταλάβω πού βρίσκεται η προσθεμένη αξία. Φυσικά δεν θα το πούμε αυτά σήμερα, αλλά ε, η μελέτη σκοπιμότητα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι επίση ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να ακούσω και τον τουρισμό περισσότερα. Τι πετύχαμε, τι καταφέραμε κλπ. Αυτά είναι τα ερωτήματα προ το παρόν. Αναγνωρίζοντα βεβαίω ότι δεν θα έχουμε χρόνο να το πούμε όλα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Σαν, λέει η κυρία Χούμπνερ. Στρέφαμε προ την Επιτροπή, την Κομισιόν, που δρομολόγησε, κατέστρεψε αυτήν την στρατηγική και ξαφνικά α, δεν έχουμε ακούσει κάτι από την Κομισιόν. Πείτε μα λίγα πράγματα, πώ βλέπει η Κομισιόν το θέμα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, άκουσα πολύ προσεκτικά τις εισηγήσεις και τον διάλογο. Θέλω να διατυπώσω μερικές γενικές παρατηρήσεις. Από την εμπειρία μας ε, από την έκθεση τη Βαλτική και σε συνάφεια με τις άλλες μακροπεριφέρειες όπως ο Δούνεβης, θα ήθελα να σχολιάσω αυτά τα οποία μου φαίνονται σημαντικά. Διάφοροι μιλητές είπαν ότι πρέπει η πολιτική βούληση να συνδυαστεί με τεχνικές δυνατότητες. Αυτό όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην ε, έκθεσή μας για τη στρατηγική της Βαλτικής προκύπτει σαφώς ότι σαφώς εργαζόμεθα για να διατηρήσουμε την πολιτική βούληση σε επίπεδα, αλλά αυτό πρέπει να συγκεράζεται με μια οργανωτική τεχνική υποστήριξη τη όλη προσπάθεια. Μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και θα το ξανατονίσουμε στην έκθεση για τη Βαλτική, η οποία είναι μια ανεξάρτητη έκθεση, έκθεση ανεξάρτητου φορέα που θα παρουσιάσουμε και στο Gdansk. Το θέμα δεν είναι μόνο να ξεκινούμε κάτι, αλλά και να το συνεχίζουμε. Η δεύτερη παρατηρήσή μου αφορά την ανάγκη να προσπαθήσουμε σοβαρά να προσαρμόσουμε την πολιτική στις δυνατότητες χρηματοδότησης και αντιστρόφως. Αυτό στα λόγια είναι εύκολο, πολύ δυσκολότερο όμως στην πράξη. Στη βελτική, ξέρουμε ότι απέδωσε προσπάθεια σε κάποιους τομείς, όχι όμως σε άλλους. Και για λόγους που είναι εύκολα κατανοητοί. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων, ε, είναι θέμα αδράνειας κάποιων πολιτικών συστημάτων, κάποιων διοικητικών μηχανισμών. Σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξε η προσδοκόμενη συνεργασία και συντονισμός. Πάντως προχωρούμε. Ο στόχος είναι εφικτός, αλλά χρειάζεται την προσοχή μας. Τρίτον, πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη να φροντίσουμε όχι μόνο για την γενική εικόνα, δηλαδή να προσπαθούμε γενικώ να δουλεύουμε με τρόπο συντονισμένο, αλλά πρέπει να εντοπίζουμε διαρκώς τα εμπόδια, τα σημεία συμφόρησης, γιατί οι γενικές ιδέες είναι σωστά διατυπωμένες για την βαλτική προκειμένου. Το θέμα είναι όμως η υλοποίηση. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε μία μελέτη όπου εστιάζουμε την προσοχή μας σε, για παράδειγμα, κεφάλαια κίνησης, τα οποία έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην πρόθεση των διαφορών έργων. Το θέμα λοιπόν αυτή τη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό και ίσω υπάρχουν πιο έξυπνοι τρόποι να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, ειδικά στη φάση τη εκείνη των έργων. Εν κατακλείδη, η εμπειρία τη Βαλτική μα δείχνει ότι υπάρχει όντω τα αξία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις υποδομές. Ο κ. Κέλλη ανέφερε τον τουρισμό, την εικόνα της Βαλτικής εν γέννη. Πρέπει όμως, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε στο δρόμο των επιτυχιών. Θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η εδαφική συνεργασία. Όταν δηλαδή και η διακυβέρνηση αποδίδει. Αυτό είναι για μας το μήνυμα. Να λέμε καταρχήν αυτό το οποίο θέλουμε και στη συνέχεια με τρόπο αξιόπιστο να υλοποιούμε. Θεσμούς, ε, όργανα, μηχανισμούς, έχουν εξασφαλίσει βεβαίως και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτήν την περίοδο και ίσως ε, ακόμη περισσότερο ε, στην περίοδο 13-20. Κύριε Αλφόνση, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή να κλείσουμε. Όχι, όχι. Να μην παρατηρούμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους. Θα τα ξαναπούμε όταν παρουσιαστεί το κείμενο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία κλείνουμε την συζήτηση για το σημείο 10. Οπότε ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά στους προσκεκλημένους μας. Αν έχετε υλικό ή παρουσιάσεις που μπορείτε να μας αφήσετε, ε, δώστε στη γραμματεία παρακαλώ για να τα προωθήσει στα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφοφορία. Ως συνήθως ε, ξεκινούμε με έναν έλεγχο. Βάλτε τα καρδιλάκια σας παρακαλώ στις γνωστές υποδοχές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 επαλήθευση στο ελέγχο που κάνουμε λειτουργούν όλα εντάξει. Uh, Η πρώτη ψηφοφορία αφορά την έκθεση ε, του Λάσρο Σούρι, αν την γνωμοδότηση μάλλον. Πολύ σύντομα ο εισηγητής αν θέλει να πει κάτι. Ε, στα αγγλικά ευχαριστώ. Ε, αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια ψηφοφορία που έχει καθυστερήσει αναδρομική. Τις τελευταίες μέρες η Επιτροπή προπολογισμό κατάφερε να αποφασίσει, να ψηφίσει και πολλοί ε, τα όσα προτείνουμε στη γνωμοδότησή μας εμείς είναι γεγονός. Όλες οι πιστώσεις πληρωμών που είχαν περικοπεί από το Συμβούλιο επανήλθαν σε επίπεδα σχεδίου προϋπολογισμού Υπήρχαν και προτάσεις ακόμα μεγαλύτερες, ακόμα περισσότερες που δεν εγκρίθηκαν ε, γιατί θεωρήθηκε ότι σε περιόδους λιτότητας ε, είναι ανεδαφικό να βάλουμε ποσά περισσότερα από το σχέδιο προπολογισμού που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες άλλες προτάσεις μειώνουν τις πληρωμές Και αυτέ επίση τι απέρριψε η συντριπτική πλειοψηφία της Επιτροπής Προπολογισμών. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπε προτάσει. εγκρίθηκαν, εκτός από μία εκ των τριών που πρότειναν οι πράσινοι, αλλά τα υπόλοιπα και τα πιλωτικά προγράμματα τα υποστηρίζει η Επιτροπή Προπολογισμών. Θα παρακαλούσα του συναδέλφου που είναι μέλη της Επιτροπής εδώ της Περιφερειακής να ψηφίσουν τα όσα συστήνει η Ευρωπαϊκή προπολογισμό για την Ολομέλεια και θα έχουμε ένα καλό προϋπολογισμό ε, για το 12 και θα είναι αύξηση στις πληρωμές κατά 8,3% στην πολιτική συνοχής που είναι το υψηλότερο ε, το υψηλότερο ποσοστό αύξηση σε όλο τον προπολογισμό. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρο, ψηφίζουμε η τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Who is against, abstain... Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Οι 5 και 6 μαζί υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. The vote is closed and it's adopted Πέρας εγκρίνεται 41 υπέρ συγχαρητήρια και πάμε παρακάτω. Στο 12. Η έκθεση της κυρίας Βέσφαλ για τη δημογραφία. Δημογραφική αλλαγή. Θέλει το λόγο η συγγήτρια. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει που λέει και η παροιμία. Τέσσερις απόπειρε χρειάστηκαν για να φτάσουμε να ψηφίσουμε επιτέλους την έκθεση για τη δημογραφική αλλαγή. Μερικοί γεράσαμε σε αυτή την προσπάθεια. Σπίσαν τα μαλλιά μας, μερικοί βγαίνουν και στη σύνταξη. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές για την πάρα πολύ καλή συνεργασία και κυρίως την επικοδομητική. Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες και κυρίως τον Χριστιαν Σοπέ και τους άλλους που συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω σήμερα να ψηφίσουμε μια έκθεση καλή όσο και ρίξει και αλευθή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Θα είπαμε από χτε ότι λυπόμαστε που φεύγει ο Σοπέ, Χριστιαν. Ε, λοιπόν, αρχίζουμε. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται σαφώς 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος γιατί 17 ηλεκτρονικά και γρήγορα αρχίζει η ψηφοφορία The vote is closed and it's adopted. Mhm. We Πέρασε. There is a, sorry, there is a oral amendment. Ε, έχουμε προφορική του κυρίου Πόγκα. Υπέρ, κατά. Όχι. Ψηφίζουμε την 21 υπέρ, όπως τροποποιήθηκε με την προφορική. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας γιατί δεν σας βλέπω. Βλέπω τον συντονιστή να κουνάει χέρι, αλλά σας όχι. Ε, κατά. Τώρα χρειάζεται έλεγχο. Τι να πάμε, δεν σηκώνετε χέρια. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 21 όπως τροποποιήθηκε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Αποχές 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται όπως και 26, 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 35 είπε. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά χρειάζεται έλεγχος για την 35 γιατί δεν ψηφίζεται. Αρχή ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Και πάλι ε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά T34. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν σηκώνουν όλα τα χέρια τους και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πέρασε, εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Απόχες, εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Απόχες, εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ Α, έχουμε μια προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανεί με την προφορική. Όχι, την ψηφίζουμε έτσι. 41 υπέρ, όπω τροποποιήθηκε. Κατά. Αποχέ. Έλεγχο. Vote open. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Sorry. Compromise 6 in favor. Υπέρ της 6 συμβαστικής κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και το δεύτερο υπέρ κατά και πάλι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 58 ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 23-21 Η 59 ήταν, όχι, το δεύτερο τμήμα της 58, Η 59 υπέρ, υπέρ της 59 κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 64. Αρχής πληροφορία. The vote is closed. And this is adopted quite large. Ε, εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 υπέρ, κατά, απόχες. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά, απόχες. Απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 με προφορική τροπολογία Γκαρσία Πέρες διαφωνεί κανείς όχι, ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε υπέρ, 77, κατά. Έλεγχος για την 77 αρχίζει τώρα παρακαλώ. Πέρας. Καταψηφίζεται. Η σημαστική 10 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, όχι, όχι, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 ψηφίπε. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω δεν ξέρω ας την ελέγξουμε την 92 αρχίζει το ηλεκτρονική ψηφοφορία Λάμπερ την 92 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται Πάμε στο συμβασμό 12. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 πε Κατά. Απορρίπτεται. Όχι, έλεγχος. Για να δούμε τι γίνεται με την 101. Ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 ψηφιπέ Κατά. Και εδώ θέλει έλεγχο συμβιβασμό. Πρώτη φορά στην ιστορία του συμβιβασμού που είμαστε τόσο διχασμένοι. The vote closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην 112 και 13 μαζί. είπε, Κατά. Απορρίπτεται. Από, α, αποχές ξέχασα, εντάξει. 114 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 και 118 μαζί είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Ξανά ηλεκτρονικά για το συμβιβασμό 14. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Θα την ελέγξουμε. Αρχή ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 και 140 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την 153 αρχής ψηφοφορία Ah, one uh, socialist Ένας νομίζω. Αποφασίστε ποιο δεν θα ψηφίζει γιατί έχετε έναν υπεράριθμο. Μεταξύ σα εν πάση περιπτώσει. Βγάλτε ένα σοσιαλιστή. So we Αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Δεν ξέρω τι ψήφισε Βίκτορ, πάντω εγκρίθηκε. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ Κατά. Να το ελέγξουμε. Το 158. Παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίψετε 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται σαφώς. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 161. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Σύμβαση 17 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168 Ειπέ. κατά αποχές εγκρίνεται 169 Ειπέ. κατά αποχές εγκρίνεται 170 Ειπέ. κατά αποχές εγκρίνεται Αιτιολογικές σκέψεις 1 Ειπέ. Abstentions, Αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά Παρακαλώ να το ελέγξουμε. για την 6 ψηφίζουμε αρχίζει τώρα η ψηφοφόρια. Πέρασε. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 με προφορική τροπολογία διαφωνεί κανείς με την προφορική όχι ωραία την ψηφίζουμε αποστροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά Μάλλον απορρίπτεται, αλλά χρειάζεται έλεγχο γιατί δεν κατάλαβα. Τη 10 ψηφίζουμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στις... Ε, προτάσεις της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Υπέρ της 1 κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σύσταση 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η σύσταση 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η σύσταση 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 6 υπέρ. Κατά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 κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 πρέπει να την ψηφίσουμε αυτή τη σύσταση Compromise Yes, it was. Η συμβιβαστική τροπολογία 13 εγκρίθηκε, έτσι δεν είναι, οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 22. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε και την 30 ακόμα σύσταση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στη στάση Επιτροπής Γυναικών. Αμπλόκ φωνάζουν από κάτω. Ναι, θα μπορούσαμε. Είστε βεβαίοι. What, Θέλετε να ψηφίσουμε ομού, αν διαφωνεί κανείς, ψηφίζουμε όλες μαζί. Τις συστάσεις Επιτροπής Γυναικών. Κανείς δεν διαφωνεί. Αμπλόκ, λοιπόν. Υπέρ. Κατά είμαστε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο. Το σχέδιο τώρα της έκθεσης ηλεκτρονικά παρακαλώ όπως τροποποιήθηκε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται. How to... Yeah, okay. So the vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 36 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια Κέρστεν. Επόμενο θέμα. Χάρτης πορείας για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Είναι γνωμοδότηση του κυρίου Ολενίτσακ. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 2-3 μαζί υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί των τροπολογιών 2-3. Σας το ξαναλέω, βλέπω μόνο χέρια σηκωμένα από τους συντονιστές. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 21 κατά. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται νομίζω, ε. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά. Γρήγορη ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24, προφορική τροπολογία, 24 με προφορική τροπολογία, υπάρχει κανείς κατά της προφορικής, όχι, επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 33 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στο σημείο 14 της κυρίας Λένα Κολάρσκα-Μπομπίνσκα. Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Δεν ξέρω αν θέλει και η κυρία Μπομπίνσκα να πάρει το λόγο. Όχι. Α, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Είναι ψηφοφορία. Α, δεν έχω ξυπνήσει καλά ακόμα. Oh, ναι, να Α, ναι, να πούμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Αλλά έπρεπε ίσως να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 50 για αυτόν. Να πάει στην ε, ε, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, ναι, σαν συντονιστής έπρεπε να είχατε υποβάλει σχετικό αίτημα. Ναι, αλλά ξέρετε αυτό επηρεάζει τη δική μας ψηφοφορία. Τέλος πάντων, θα ψηφίσουμε. Εγώ, αν μου κάνει, μου υποβάλλετε το αίτημα, το μεταφέρω. Τροπολογία, συμφασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 Τροπολογία 7 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22, τροπολογία 22, με προφορική τροπολογία. Κάποιος αντιτίθεται στην προφορική τροπολογία, όχι. Επομένως προχωρούμε στην τροπολογία 22, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τελική ψηφοφορία, η ηλεκτρονικής ψηφοφορίας άρχεται. Πέρας. Έχουμε 40 ψήφους υπέρ και συγχαίρουμε βεβαίως τη συνάδελφο κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τροπολογίες που υποβάλλατε, για την συνεργασία, ε, το γεγονός ευχαριστώ τους, ε, συγγνώμη, τους ε, για την ε, καλή συνεργασία. Πάρα πολύ ωραία λέει η πρόεδρος. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Τι κάναμε, το εγκρίναμε ήδη. Α, ωραία. Άρα είμαστε τώρα έτοιμοι για τον Γενικό Διευθυντή κύριο Dirk Άνερ, ο οποίος όμως έχει καθυστερήσει είναι αργοπορημένος. Και επομένως θα μπορούσαμε να περάσουμε στο σημείο 17. Έχουμε όλους όσους πρέπει να είναι εδώ. Όχι. Uh, so we, we adopt this change, no, no. Hmm? So we, we change. I say it, no. Yeah, we will Dear colleagues, as Madame Constance Krell is not here with. Η κυρία Κωνσταντίνα Κρόλ δεν είναι μαζί μα, άρα το σημείο 17 που αφορά έκθεση σχετικά με την επίσκεψη τη αντιπροσωπεία Ρέτζι στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα μα απασχολήσει την επόμενη φορά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τη απουσία τη, αν είναι δυνατόν. Επομένως, τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη πριν από το μεσημερινό διάλειμμα είναι αυτό της ανταλλαγής απόψεων με τον κύριο Ντίρκ Άχνερ θα ήθελα να σταματήσουμε για λίγο. Θέλω να πω να μην εγκαταλείψετε όμως την αίθουσα. Ένα ευέλικτο διάλειμμα, λέει η Πρόεδρος, θα κάνουμε. Σε πέντε λεπτάκια θα έρθει, είναι καθοδόν, το έχουμε ελέγξει.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 μην ξένα δεν βλέπω ότι ο Dear colleagues, I hope that uh, we, we can start, restart our uh, meeting. We... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε και πάλι. Δίνω τον λόγο αμέσω στον Γενικό Διευθυντή Κάνα, ο οποίο ε, θα μα παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας που ενέκρινε χθε η Κομισιόν όσον αφορά την άλυση των ε, σφαλμάτων στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή και τις ε, σχετικές δράσεις που έχει αναλάβει στο Ρεκομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά η κυκλοφορία ήταν απίστευτη στην περιοχή. Κάθε χρόνο συζητούμε την κανονικότητα των στοιχείων και τα ασφάλματα στην εκτέλεση του κοινοτικού προπολογισμού. Κάθε χρόνο διαπιστώνουμε στο τέλος ότι στην πολιτική συνοχή και δι στον ομέα της περιφερειακής πολιτικής παρισφύουν σφάλματα. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Και αυτό προκύπτει από τις συγκρίσεις με το προηγούμενο έτος. Με βάση λοιπόν την εμπειρία των τεσσάρων τελευταίων ετών, δηλαδή από το 2007 ως σήμερα, αναλύσαμε τα σφάλματα και προσπαθήσαμε να συναγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα, για τα μαθήματα, τα συμπεράσματα, αν θέλετε, που συναγάγαμε βάσει αυτής της ανάλυσης. Η βάση δεν είναι μόνο η δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου. Χρησιμοποίησαμε και δύο άλλες βάσεις. Η μία είναι η εργασία των υπηρεσιών της Κομισιόν. Και προκειμένου έχουμε εδώ στοιχεία 5 ετών. Και έχουμε βεβαίως και την συνεισφορά των εθνικών αρχών, των εθνικών ελεγκτικών αρχών, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικά επάλληλα επίπεδα ελέγχου, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα συνδιαχείρισης. Όλα τα επίπεδα ελέγχου διαδραματίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο. Συνεπώ, ας δούμε τα γενικά καταρχήν αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ την κατάσταση βάσει της ανάλυσης του ελεγκτικού συνεδρίου για την περίοδο 2006-2009. Δύο είναι τα μηνύματα από το Ελληνικό Συνέδριο. Το πρώτο αφορά τη συχνότητα των ελέγχων ή μάλλον των σφαλμάτων κατά τη των ελέγχων και το δεύτερο είναι ο υπολογισμό, η μπλε γραμμή με τον αριθμό των σφαλμάτων. Χαιρόμαστε πολύ, διότι το 2009 η μπλε γραμμή, όπως είδατε, έχει κατέβει πάρα πολύ. Το 2009 ήταν από πολλές απόψεις μια ειδική χρονιά, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Με την έννοια ότι για την περίοδο 2007-2013 ιδιαίτερα υψηλά ποσά πληρωμών έγιναν μέσα σε ένα χρόνο στα κρατη Το 2009 λοιπόν είχε συγκεντρωμένες πολλές πληρωμές. Μάλιστα εκεί προσθέθηκαν και προγράμματα από την περίοδο μέχρι το 2006. Οπότε για φέτος με βάση αυτά εκτιμούμε ότι ο αριθμός των σφαλμάτων θα διακυμανθεί και πάλι, αλλά ότι εν γέννη η συνότητα θα συνεχίσει να πέφτει σε σχέση με τα έτη 2006 και 2007. Γιατί? Διότι αναλάβαμε σημαντικές δράσεις, λάβαμε μέτρα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι για την περίοδο 7-13 πολλοί κανόνες τροποποιήθηκαν ακριβώς για να μειώσουμε, για να μειωθεί ο αριθμός των σφαλμάτων. Ας αναλύσουμε μαζί τώρα τα σφάλματα και ας πούμε δύο λόγια για τα μέτρα τα οποία έλαβε η Κομισιόν. Τι είναι σφάλμα καταρχήν. Ας πάμε στην διαφάνεια υπαριθμών 6. Σφάλμα προκύπτει όταν μια συναλλαγή, μια κίνηση δεν υλοποιείται σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις με αποτέλεσμα να δηλωθεί Παρατύπω δαπάνη στην Κομισιόν. Να το πω και είναι Τι δεν είναι σφάλμα. Διότι στην κοινή γνώμη γενικώ ε, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Σφάλμα δεν σημαίνει. Σφάλμα δεν σημαίνει ότι κονδύλια εξαφανίστηκαν, χάθηκαν ή ότι σπαταλήθηκαν. Όχι, μιλούμε για περιπτώσεις όπου τα χρήματα όντως κατέληξαν στα χέρια αυτών στους οποίους είχε προβλεφθεί να καταλήξουν. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και η χρήση των κονδυλίων συνιστά παρατυπία. Παρατυπία, για παράδειγμα, στον τομέα των δημοσίων προμηθειών των δημοσίων συμβάσεων, αν θέλετε. Επειδή κάποιοι κανόνες δεν εφαρμόστηκαν ορθώς. Ή μιλάμε για παρατυπίες στην περίπτωση του ΦΠΑ ή στην ανάκτηση του ΦΠΑ. Τα κονδύλια δηλαδή απορροφήθηκαν από το έργο. Το έργο όντω υλοποιήθηκε, μπορεί να το δει κανεί εν τούτης, στις πληρωμές σημειώθηκαν παρατυπίες ε, σαν αυτές που προανέφερα. Πολύ πολύ σπάνια με τους ελέγχους που διενεργούμε αποκαλύπτουμε και περιπτώσεις απάτης. Περιπτώσεις δηλαδή όπου με δόλο συγκεκριμένα άτομα προσπάθησαν να αποσπάσουν ε, πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος τον οποίο είναι σπάνιες οι απάτες είναι ότι τα κράτη-μέλη καταρχήν προσέχουν πάρα πολύ και ότι συναφώς λαμβάνουν μέτρα με το που θα προκύψουν σχετικά υποψίες. Ο δεύτερος λόγος, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός, είναι ότι κάθε φορά που αποκαλύπτουμε μια απάτη υπάρχει καταγγελία ή έστω και υποψία απάτης, τότε αμέσως ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές. Στην Κομισιόν είναι η Όλαφ, είναι το γραφείο καταπολέμησης της απάτης και φυσικά τις αρμόδιες υπηρεσίες στο κρατός μέλος. Δρομολογείται τότε έρευνα και πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολλές τέτοιες υποθέσεις Σε πάρα πολλές ε, όμως από αυτές το τελικό έβριμα ήταν ότι δεν πρόκειται περί επάτης. Κάποιες άλλες υποθέσεις βεβαίως προχώρησαν και απαιτήθηκε να χρησιμοποιήσουμε ένδικα μέσα κατά των απαταιώνων. Πάντω παραλαμβάνω και το υπογραμμίζω ότι οι πραγματικέ περιπτώσει απάτη ω τώρα είναι πολύ λίγε. Δύο λόγια τώρα για τι μεθόδου, την μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για όλου αυτού του υπολογισμού. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι το ελεγκτικό συνέδριο χρησιμοποιεί πολύ συγκεκριμένη στατιστική μεθοδολογία όπου για κάθε συγκεκριμένη χρονιά παίρνει ένα, καταγράφει θέλετε, ένα στιγμιότυπο της κατάστασης τη συγκεκριμένη χρονιά. Αυτό είναι αρμοδιότητα ούτως ή άλλως του ελεγκτικού συνεδρίου για τους σκοπούς της δήλωσης αξιοπιστίας για το συγκεκριμένο έτος. Μία δυσκολία είναι τα πολιτική προγράμματα. Διότι αν στο έτος νη υπάρχει σφάλμα το οποίο αποκαλύπτεται το έτος N συν 1 ή N συν 2, τότε αυτομάτως πρέπει να γίνει διόρθωση αναδρομικά για το έτος n. Και τότε πρέπει να αλλάξουμε διάφορα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, για το συγκεκριμένο έτος. Πράγμα το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, δηλαδή 7 χρόνια μετά, μετά από ένα σωρό διορθώσεις, πρέπει εμείς να καταλήξουμε σε ένα συνολικό συμπέρασμα όσον αφορά τα ασφάλματα της προγραμματικής περίοδου. Αυτό δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί στη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου, έτσι όπως δουλεύει το ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς, για την περίοδο 94-95, έχουμε οριστικά στοιχεία και διαπιστώσαμε ότι μετά από όλες τις διορθώσεις, στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, ο τελικός αριθμός σφαλμάτων είναι πολύ πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το ετήσιο στιγμιότυπο, την ετήσια απογραφή, αν θέλετε, που κάνει το ελληνικό συνέδριο. Το ελληνικό συνέδριο βεβαίως ορθώς υποστηρίζει ότι ο προπολογισμός της Ένωσης είναι ούτως ή ετήσιος και ότι η ανάλυση πρέπει να είναι και αυτή ετήσια. Λοιπόν, για να έχει κανείς μια σαφή εικόνα της κατάστασης πρέπει να κάνει και τα δύο. Και αυτό που κάνει το ελληνικό συνέδριο και αυτό που κάνουμε εμείς. Έχουμε λοιπόν δύο προσεγγίσεις, μια ετήσια και μια πολυετή. Εμείς αποδεχόμεθα απολύτως πλήρω τη μεθοδολογία του ελληνικού συνεδρίου. Όμως έχουμε μια ένσταση όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων. Και προκειμένου το ελεγκτικό συνέδριο ασχολείται καταρχήν βεβαίω, όπω είπα, με το αν υπάρχει σφάλμα ή όχι. Εάν υπάρχει επίπτωση, στην περίπτωση που είναι ποσοτικοποιήσιμο το σφάλμα. Και εν συνεχεία το ελεγκτικό συνέδριο προβαίνει στην τελική του κρίση. Εμείς, στην περίπτωση ποσοτικοποιήσιμου σφάλματος, φροντίζουμε να ανακτήσουμε τα σχετικά ποσά από τις ε, αρχές του κράτους μέλους ή την διαχειριστική αρχή. Εννοείται σε αυτές τις περιπτώσεις υπερισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Εμείς πρέπει να ανακτήσουμε τους σχετικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της αναλογικότητας. Και ένα καλό παράδειγμα σχετικά είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Στον τομέα αυτών, το ελεγκτικό συνέδριο, όταν εντοπίζει σφάλμα, ε, στην περίπτωση που το σφάλμα αυτό είναι αμεληταίο, το ελληνικό συνέδριο λέει ε, ξέχνα το, αν είναι μέσα μεγέθους εκεί διαπιστώνεται ότι κάτι πήγε στραβά. 100%. Όμως όταν το σφάλμα αυτό επαναλαμβάνεται, τότε υπάρχει απώλεια για τον προϋπολογισμό και για ένα μεσοσφάλμα μπορούμε να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε 50%, 20%, 10% των σχετικών πόρων. Θέλω να πω δηλαδή ότι από ποσοτική απόψεω, όσον αφορά την αξία του σφάλματο, η γνώμη δική μα μπορεί να διείσταται σε σχέση με αυτήν του ελληνικού συνεδρίου. Δεν σημαίνει αυτό πολύ συχνά, αλλά κάθε χρόνο έχουμε μία ή δύο περιπτώσει όπου υπάρχει, υπάρχουν διστάμενε απόψει μεταξύ ελληνικού συνεδρίου και κομισιών. Α δούμε την δική μας τώρα ανάλυση και την ανάλυση του ελεγκτικού συνεδρίου και την εικόνα των διαχειριστικών ερχών. προκύπτει σαφώς ότι τα ασφάλματα συγκεντρώνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την επιλεξιμότητα. Είτε στο επίπεδο των έργων, είτε δαπανών, όπου δηλαδή αιτήσει πληρωμής υποβλήθηκαν που δεν συνάδουν με τους κανόνες μας. Η άλλη κατηγορία προβλημάτων άπτεται των δημοσίων συμβάσεων. Βλέπετε ότι ακόμη και σήμερα πολλά σφάλματα καταγράφονται ως παρατυπίες στα κρατημέλη στον τομέα αυτών. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο έκτο, βεβαίω είναι λιγότερα τα προβλήματα. Πάντω ε, να θυμίσω ότι τα περισσότερα σφάλματα προέρχονται από θέματα επιλεξιμότητα. Α δούμε όμω ε, τι επόμενε διαφάνειε. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ παρατηρούμε πρώτον ότι οι προσφορές δεν αξιολογούνται όπως θα έπρεπε. Επειδή τα κριτηρία ενδεχομένω δεν είναι σαφώς καθορισμένα ή δεν είναι καθορισμένα από την αρχή ή δεν ελήφθησαν υπόψη όπως θα έπρεπε. Το άλλο πρόβλημα που παρατηρούμε συχνά είναι η απουσία εληφθησαν υποψη οπω θα επρεπε το αλλο προβλημα ή μιας ορθά κατακτισμένη σύμβασης. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά και δει όταν τρέχει ένα μεγάλο έργο. Με το που θα εμφανιστεί ένα πρόβλημα, θα περιθουν έργα ή τροποποίηση κάποιου αντικειμένου. Η τάση, όπως καταλαβαίνετε, και είναι φυσικό αυτό, είναι να πει ο κύριος του έργου, συνεχίζω με τον ανάδοχο που γνωρίζω, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τα μηχανήματα στο εργοτάξιο, ας συνεχίσουν να κάνουν και το συμπληρωματικό έργο. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες της σχετική οδηγίας περί δημοσίων συμβάσεων απαιτούν σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση πάνω από κάποιο όριο βεβαίως, να προκηρυχθεί ξεχωριστός νέος διαγωνισμός. Και αυτό είναι, όπως είπα, ένα από τα προβλήματα που ανακύπτουν συχνά. Πολλέ φορές έχουμε προβλήματα ως προς τις απαιτήσει δημοσιότητες. Δεν αρκεί η δημοσίευση ενός διαγωνισμού στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου. Η ανακοίνωση ανακοίνωση πέρι της μελλοντικής ανακοίνωσης του διαγωνισμού. Πολλές φορές αυτοί οι κανόνες, αυτές οι ελάχιστες απαιτήσει δεν τηρούνται. Αν έρθουμε τώρα στους κανόνες επιλεξιμότητας, ένα από τα σφάλματα τα οποία οδηγούν σε μη ανακτήσιμους πόρους, Ανοίξω σε αυτήν την κατηγορία. Πολλές φορές έχουν γίνει λάθη στο ποσοστό συγχρηματοδότησης ή στην ε, ανάκτηση του ΦΠΑ. Κάτι το οποίο εμένα προσωπικώς με ανισχύει πολύ, όπως και του συνεργάτες μου, είναι τα λεγόμενα αναδρομικά έργα. Και επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω εντάχει τι είναι αυτό το πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της περίοδου υλοποίησης ενός προγράμματος, ενδέχεται, και εν μέρει επιτρέπεται, ενδέχεται όμως ένα κράτος μέλος να επαρέλθει σε υλοποιηθέν έργο από το παρελθόν που έχει υλοποιηθεί με εθνικούς πόρους και το έργο αυτό να προσπαθήσει να το εντάξει έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί με νέους πόρους. Εμένα πρέπει να σας πω προσωπικά αυτή η πρακτική δεν μου αρέσει γιατί προκαλεί δύο κατηγορίες προβλημάτων. Πρώτον, έχουμε το θέμα της προσθετικότητας και δεύτερον, πολλές φορές το έργο ακριβώς επειδή είχε υλοποιηθεί μόνο με εθνικούς πόρους και είχε σαφώς εξεταστεί, δεν επανεξετάζεται αυστηρά με τους νέους κανόνες, τους κοινωτικούς κανόνες. Και υπάρχουν περιπτώσεις, όπως φαντάζεστε, όπου οι εθνικοί κανόνες είναι πολύ πιο χαλαροί σε σχέση με τους κοινωτικούς. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι ανεκτό σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ανεκτό ή συμβατό με τους κοινωτικούς κανόνες. Και αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε και φέτος αρκετές φορές πρέπει να πω. Πρόκειται για πρόβλημα το οποίο θα ήθελα πραγματικά να συζητήσω μαζί σας στο πλαίσιο της συζήτησης για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ένα άλλο ζήτημα είναι η γεωγραφική κατανομή των σφαλμάτων. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο συγκεκριμένες χώρες εμφανίζουν τον υψηλότερο αριθμό, του υψηλότερο πλήθος σφαλμάτων. Αν δούμε τις δύο-τρεις χειρότερες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν ταυτόχρονα και τα δύο τρίτα των σφαλμάτων που εντοπίζουμε σε ένα χρόνο. Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο την ετήσια εικόνα, αλλά μια πιο απλωμένη εικόνα σε 4-5 χρόνια. Να δούμε εάν η εικόνα αλλάζει ουσιαστικά από τη μία χρονιά στην άλλη, πράγμα το οποίο θα μας έκανε να σκεφτούμε ότι υπάρχει κάποιο συστημικό πρόβλημα. Το κάναμε λοιπόν αυτό και διαπιστώσαμε όντως ότι στην Ισπανία και στην Ιταλία έχουμε τα περισσότερα σφάλματα συστηματικά θα έλεγα. Μάλιστα θα ήταν δικό να πω ότι αφορά αυτό όλη τη χώρα, αλλά αφορά συγκεκριμένες περιφέρειες. Και εκεί έχουμε δραστηριοποιηθεί, έχουμε έρθει σε επαφή με τις ε, εθνικές και τοπικές αρχές για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να λύσουμε το πρόβλημα. Το οποίο με οδηγεί στο τι κάνει η Κομισιόν τώρα κάθε χρόνο με τη μορφή ελέγχων όλων των πληροφοριών που παίρνουμε από επιχειρησιακή απόψεω. Αν δούμε λοιπόν τα 300 τόσα προγράμματα, 340 προγράμματα που έχουμε περίπου, αν τα δούμε όλα αυτά, θα έλεγα ότι στο 90% με βάση τα στοιχεία από τους μου και τα στοιχεία των αρχών παρακολούθησης. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι αρκετά αξιόπιστα. Το θέμα λοιπόν είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 10%. Στην περίπτωση των συναδέλφων του Κοινωνικού Ταμείου, οι αριθμοί είναι λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα. Προσπαθούμε λοιπόν, κάθε φορά που εντοπίζουμε τέτοιου είδου προβλήματα, να εισάγουμε μια επιφύλαξη στην ετήσια έκθεσή μας, ενώ παραλαβαίως προσπαθούμε να κάνουμε κάτι με τις υπηρεσίε μας και τις αρχές του κρατούς μέλους. Αν δούμε το 2010, θα έλεγα ότι τα περισσότερα προβλήματα που οδήγησαν σε δήλωση επιφύλαξης θα μπορούσαν σύντομα να επιληθούν σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Και ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η συνεργασία με τα περισσότερα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες αντιστοίχως βελτιώνεται συνεχώς. Κάτι το οποίο μας βοηθάει πολύ να επιλύουμε τα προβλήματα. Δύο πράγματα κάνουμε για να λύσουμε τις δύο κατηγορίες προβλημάτων. Πρώτον, επεμβαίνουμε προληπτικά. πως ξέρετε υπάρχουν επιτροπές παρακολούθησης. Ε, συστούμε ένα δείγμα προγραμμάτων. Εμείς είμαστε παρατηρητές, έχουμε εμπειρογνώμονες και μπορούμε να πιστήσουμε την προσοχή των στελεχών των επιτροπών παρακολούθηση στα προβλήματα τα οποία εντοπίζουμε. Έχουμε αιτήσεις συσκέψεις με τις διαχειριστικέ αρχές και τις αρχές ελέγχου, όπου συζητούμε συγκεκριμένα τα προβλήματα που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτου και ζητούμε σχετικέ λύσει. Και τρίτον, προσπαθούμε είτε σε πολυμερή είτε σε διμερή βάση να παρέχουμε διαρκώς κατευθυντήριε γραμμές στις διαχειριστικές και ελληνικέ αρχές στα κρατημέλη. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η προληπτική δράση θα αποτελέσει σημαντική πρόοδο. Φυσικά υπάρχει και η διορθωτική δράση, υπάρχουν διορθωτικές ενέργειες, όπου πρέπει να σας πω είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά την διακοπή, για παράδειγμα, των πληρωμών. Διακοπή ή αναστολή πληρωμών. Αν εντοπίσουμε πρόβλημα, προτιμούμε να καθίσουμε κάτω με το κράτος μέλος, να αναστείλουμε, από είπα, τις πληρωμές και μετά να τις επαναφέρουμε αν όλα πάνε καλά. Αν και ένας χρόνος συστηματικών ελέγχων δεν είναι επαρκής για τη συναγωγή γενικών συμπερασμάτων. Θα έλεγα ότι η υποδοχή που είχαμε από τα κρατημέλη ήταν εξαιρετικά καλή στην προσεγγίση μας αυτή. Σε άλλες ε, περιπτώσεις, όπως είχατε προτείνει και εσείς, εστιάζουμε την προσοχή μας στις περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι ολοχεύουν μεγαλύτερη κίνδυνη λόγω ενδεχομένω του ύψου των κονδυλίων ή λόγω του ιστορικού. Σε χώρες περιφέρειες ε, όπου οι ελληνικές αρχές δεν κάνουν ακόμη επαρκώς τη δουλειά τους. Πρέπει να σας πω παραδότη το 70% των ελεγκτικών αρχών με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Το 1 τρίτο χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. Όταν λοιπόν πάρουμε τα αποτελέσματα του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και τα δικά μας εννοείται, εμείς δίνουμε συνέχεια στα ευρήματα για να επανέλθω στις δημόσιες συμβάσεις και το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για την ανάλυση των σφαλμάτων, διοργανώνουμε σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις κλπ. για να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν πλήρως το κοινοτικό δίκαιο. Όσον αφορά την επιλεξιμότητα, για αυτήν την περίοδο ξεκινήσαμε και θα το κάνουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον να χρησιμοποιούμε την προσέγγιση των απλουστευμένων στοιχείων κόστους. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα απλοποιημένα κόστη και χαίρομαι γι' αυτό. Ελπίζω μάλιστα ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο με τη μέθοδο αυτή του απλουστευμένου κόστου, θα έχουμε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά ειδικά σφάλματα, τα αναδρομικό συνταχθέντα έργα, έχουμε στείλει κατευθυντήριες γραμμές στις διαχειριστικές αρχές και όσον αφορά την ειχνηλάτηση των ε, συναλλαγών. Έχουμε κλείσει εν μέρη την περίοδο 7-13 και έχουμε επενδύσει τους τελευταίους μήνες πολύ σε δουλειά, σε χρηματοοικονομικές τεχνικές που είναι ένα νέο εργαλείο μάλλον ένα εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιείται εκτεραμένα, για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε, να χειριστούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Ενώ τώρα της προγραμματικής περίοδου 2014-2020 ο Επίτροπος θα είναι μαζί σας το απόγευμα να σας πει δύο λόγια. Το μήνυμά μας είναι ότι θα συνεχίσουμε υπέρ της περαιτέρω απλούστευσης. Οι έλεγχοι θα βασίζονται στον κίνδυνο. Θα συνεργαστούμε στενότερα με τις αρχές ελέγχου και ειδικά με αυτές που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Θα προσπαθήσουμε επίση να πλουστεύσουμε τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εν γέννη και θα προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε ένα σύστημα, έναν ε, μηχανισμό που δανειστήκαμε από, τη, από το χώρο της γεωργίας για να καθιερώσουμε μια ετήσια διαδικασία καθάρισης πληρωμών προσαρμοσμένη φυσικά στη συνοχή. Αυτή η ετήσια διαδικασία καθάριση θα γλιτώσει και εμάς και τα κρατημέλη και τους δικαιούχους από την διαρκή συσσόρευση προβλημάτων επί 7 χρόνια αποτέλεσμα να μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνο στο τέλος της προγραμματικής περίοδου με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτή είναι λοιπόν η νέα μας προσέγγιση. Εν κατακλείδη να πω ότι πρώτον Έχουμε τη χαρά να έχουμε πίσω μας εμπειρία 4-5 ετών, εμπειρίες και στοιχείων. Να σας ευχαριστήσω επιπλέον διότι χάρη και στις δικές σας προσπάθειες το πλήθος των σφαλμάτων και η συνότητα των σφαλμάτων έχει μειωθεί θεαματικά. Είναι σήμερα κατά το μισό του ποσοστού που είχαμε στο παρελθόν, μείωση μεγαλύτερη από 50% και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχίσουμε να μειώνουμε τα σφάλματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα θεωρούμε πάντα το ποσοστό αυτό υψηλό. Ιδιαίτερα στην περιφερειακή πολιτική, στο ΕΚΤ, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λόγω ακριβώς της φύσης των πληρωμών του ΕΚΤ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και εκεί σημειώσαμε ταχύτατη πρόοδο. Μειώσαμε και εκεί πολύ τα σφάλματα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να βελτιώνουμε το σύστημα στο μέλλον. Μάθαμε πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία. ως το τέλος του 2005 15 όταν θα γίνονται και οι τελευταίες πληρωμές για αυτήν την προγραμματική περίοδο. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν ακόμη περισσότερο τα συμπεράσματα αυτά εν ώψη του νέου κανονισμού ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να είναι ακόμη πιο αποδοτικό. Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να κλείσω χωρίς να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιστροπής σας για την υποστήριξη μας που όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά που συζητούσαμε όλα αυτά τα καθόδη πολύπλοκα θέματα. Ήταν πολύπλοκα και ακαθόδη. Και αυτό φαίνεται και από το ότι η εξοπιστία τη εν γέννη πολιτικής μας εξαρτάται από αυτά. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κάποιος να κάνει σχόλια, να υποβάλει ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άννα. Λέει ο κύριος Γκάιερ. Χαίρομαι που σας ακούω εδώ, αν και είμαι ένα αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι στην Επιτροπή, γιατί αυτά που μας λέτε είναι καθημερινή δουλειά ψωμοτήρη για μας σε αυτή την Επιτροπή. Πώς ε, μπορούμε να μειώσουμε τα ποσοστά σφάλματος. Ε, μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Συμφωνούμε ότι το θέμα των σφαλμάτων σε πληρωμές για τα περιφερειακά ταμεία είναι και ένα θέμα που αφορά την ακαιρεότητα και των θεσμικών οργάνων και πολλές φορές τη διακυβεύει και την υπονομεύει. αυτό θέλουμε να μειωθεί και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Η σε έκθεση του Ελεκτικού συνεδρίου πέρυσι για το έτος 2009 διαπίστωσε μείωση στο μισό των σφαλμάτων. Είχαμε ένα ποσοστό 11% στις πληρωμές στο παρελθόν και το 2009 σε αυτό το κεφάλαιο που δεν καλύπτει με μόνο την περιφερειακή πολιτική στο ελεγκτικό συνέδριο, αλλά ευρύτερα θέματα, τελικά έφτασε να είναι στο μισό περίπου το ποσοστό. Βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Και ως σκιώδης εισηγητής για την απαλλαγή της Επιτροπής για το έτος 2010, θα ήθελα να σας αποσπάσω μία εκτίμηση ε, και μία πρόβλεψη. Περιμένετε να πέσει αυτό το σφάλμα κάτω του 5%. Ε, σύμφωνα με τα όσα ζητεί και το ελεκτικό συνέδριο και έχω δύο συγκεκριμένες τεχνικές ερωτήσεις. Μιλήσατε για την ε, επιστροφή των χρημάτων και την επανίσπραξη. Δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό καν αλλά αν έχει διαπιστωθεί μια εσφαλμένη πληρωμή και διορθώνεται με επανακαταβολή του ποσού, το σφάλμα αυτό έρεται, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό το σφάλμα που ήρθε, ήρθε, καταγράφεται πουθενά, προσμετράτε εκ των υστέρων. Μετά την επανάκτηση της πληρωμής διορθώνεται αυτό όταν κλείσουν οι λογαριασμοί ή το μετράμε με διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να το συζητήσω αυτό και με το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί εκείνοι λέγουν ότι είναι δύο δυνατότητες ε, να αποφευθεί ένα σφάλμα. Ε, είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων. Είτε το αποφεύγεις είτε το διορθώνεις. Άρα όταν το διορθώνεις, για να το βρεις το έχεις μετρήσει. Μετά δεν θα πρέπει να το ελέγξουμε και να κάνουμε μια επαλήθευση, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον θα έπρεπε να, γίνει και να διορθωθεί. Και το δεύτερο, ναι, οι διακοπές, οι αναστολές. Εμείς που ελέγχουμε τον προϋπολογισμό, χαρήκαμε όταν ακούσαμε αυτά που μας είπαν συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Γιατί στην τελευταία της έκθεση είχαν πάρα πολύ συνεπή στάση και διέκοπταν τα επιχειρησιακά ε, σχέδια όταν έβλεπαν ότι υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό και μειώθηκε τόσο πολύ το σφάλμα στο κοινωνικό ταμείο. Και ήταν στο, στο πράσινο πεδίο, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του ελεγκτικού συνεδρίου, δηλαδή κάτω από το 2%. Τεράστια επιτυχία. Αυτό το μέσο εσείς το χρησιμοποιείτε με κάποιο τρόπο, με την ίδια ένταση όπως και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και πόσα προγράμματα έχετε να στείλει αυτό το καιρό. Thank you and Lambert Van Ευχαριστώ, Lambert Van Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για την έκθεσή σα Είναι και αυτή η αιτήσια για την εξέλιξη κάθε φορά. Καλό είναι για να δούμε τους νέους κανονισμούς, πώς θα διαμορφωθούν και πώς αυτές οι απαιτήσει θα μεταφραστούν στη νέα προγραμματική περίοδο. Πάντως ε, προσωρινά αφορά την τρέχουσα περίοδο. Χαίρομαι και εγώ και συμφωνώ, όπως ο κύριος Γκάιερ, για τις ουσιαστικές βελτιώσεις. Ε, αν δούμε και σε σχέση με την περσινή κατάσταση, ε, τα αιτήσια στοιχεία και οι αριθμοί εκτείνονται και κυμαίνονται ε, με την πάροδο των ετών βελτιώνεται εντάξει η κατάσταση αλλά δεν παραμένει σταθερή. Έχει καμπανεβάσματα. Την επόμενη φορά μπορεί να έχουμε άλλα στοιχεία ε, με ε, χώρες έτσι, και γεωγραφική κατανομή επηρεασμένη από διάφορους παράγοντες και να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι για την έκθεση. Η ερώτησή μου ε, πηγαίνει προς τη συγχρηματοδότηση πάντα είναι ή συνυπευθυνότητα ή συγχρηματοδότηση, ξέρω εγώ μέχρι 50% αν είναι για το κοινωνικό ταμείο ή λίγο χαμηλότερη, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξετε περισσότερο προς την κατεύθυνση της ευθύνης των κρατών μελών και να τις αναλαμβάνουν και εκείνοι οι εθνικές ε, ε, δηλώσεις διαχείρισης Ε, θα πρέπει να βαραίνουν τα κράτη, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την αποκεντρωμένη διαχείριση και να είναι και υπόλογα. Προσωπικά είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Το έχω ξαναπεί και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και το ζήτησα, αλλά δεν με ικανοποιεί η ταχύτητα με την οποία προχωράει το θέμα. Το ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Άνερ, θα βοηθούσε στη συζήτηση που γίνεται αυτό τον καιρό να κάνουμε κανένα βηματάκι προς τα εμπρός. Δεύτερη παρατηρήση. Κοιτάω δεξιά και αριστερά. Και βλέπω ότι μιλάτε για τα καπολέμηση παρατυπιών, λαθών κτλ. Όλα αυτά οδηγούν σε περισσότερους εθνικούς ελέγχους και εθνική δραστηριότητα. Και ο αριθμός των ελέγχων που είναι αλλεπάλληλοι ε, είναι πολύ, γιατί συνήθως υπάρχει αρχή ε, το ένα πρόγραμμα, ένας λογιστικός έλεγχος. Αλλά αυτό έχει ξυλωθεί. Καμία φορά έχουμε και 14 ελέγχους, καλά υπερβάλλω, 7 ας πούμε, αλλά όχι έναν. Στο εσωτερικό των κρατών μελών πριν φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε σε θέση να μειώσουμε ε, αυτά σε απλά προγράμματα, ε, αυτά, τα διάφορα στρώματα και επίπεδα διαδοχικών λογιστικών ελέγχων και κάτι άλλο που επίσης είπα στην Επιτροπή Ελέγχου, τον προϋπολογισμό, γίνεται λόγος και θα ψηφίσουμε για τον νέο χρηματο... Μάλλον δημοσιονομικό κανονισμό και ε, σε πολλούς τομείς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γίνεται λόγο και το είπατε και εσείς, για καινοτόμε μορφές χρηματοδότησης, ανάληψη κινδύνου, δυνατότητες, δάνεια κτλ. Θα τα κοιτάξουμε αν μπορεί να γίνει και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Καταλαβαίνετε, και εγώ καταλαβαίνω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τριπλασιάσει ή να τέτραπλασιάσει αυτού του είδους τα μέσα την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό γιατί αν ε, επεμβαίνει και η τράπεζα θα έρθουν και τράπεζες οι οποίες ε, δεν είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν και τις προσελκύουμε ε, να μπουν σε τέτοια προγράμματα όταν υπάρχει και η τράπεζα επενδύσεων. Ωραία. Τι γίνεται όμως με το σύστημα ελέγχου. Αν είναι τόσο υπερβολικό και επιβαρημένο δεν ξέρω λειτουργήσει. Δηλαδή να μην μας παρασύρει ο ενθουσιασμός και η χαρά μας για τα καινοτόμα μέσα και να μην ε, αποδειχτεί αυτό τροχοπέδι τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Και δεν πάμε τόσο καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση αυτή. Θα την αξιοποιήσουμε, θα τη χρησιμοποιήσουμε πολύ και θα είμαστε σε επαφή με τις υπηρεσίες σας στην νομοθετική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρακάκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άννα για το γεγονός ότι είναι σήμερα μαζί μας και μας έκανε μια τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ανάλυση της έκθεσης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής για την έγκαιρη, ξεκάθαρη και εξαιρετικά κατατοπιστική ανάλυση των λαθών στην πολιτική συνοχής. Είναι αδιαφεσβήτητο ότι μόνο όταν γνωρίζουμε πού κυρίω γίνονται τα λάθη θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και ή δυνατόν να τα μηδενίσουμε στο μέλλον. Όπως προκύπτει από τη σημερινή παρουσίαση του κυρίου Άνερ, η πλειοψηφία των προγραμμάτων υλοποιείται χωρίς σημαντικά λάθη, κάτι που θα πρέπει να μας κάνει να αξιολογήσουμε σε άλλη βάση το γεγονός ότι αναρρύθμιτες συζητήσεις αφιερώνονται κάθε χρόνο στα λάθη και τις παρατυπίες της πολιτικής συνοχής. Ως μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού θα ήθελα να τονίσω ότι πολλές φορές στις συνεδριάσεις μας διατυπώνονται εξαιρετικά αρνητικά σχόλια για την πολιτική συνοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να έρθετε κύριε Άνερ και στην Ελόγω Επιτροπή προκειμένου να αποκαταστήσετε την εικόνα της πολιτικής με βάση τα νέα δεδομένα. Το κύριο ερώτημα που προκύπτει κατά τη γνώμη μου είναι με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι όλα τα προγράμματα θα παρουσιάζουν το βέλτιστο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας. Είναι ξεκάθαρο ότι λαμβάνονται πλέον τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα λάθη που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα, ενώ τα λάθη που σχετίζονται με τη διαδικασία ελέγχου δεν αποτελούν πλέον κύρια παράμετρο του λαθών. Ωστόσο, ακόμη και αν τα λάθη που σχετίζονται με την πολιτική συνοχή μηδενιστούν, οι δημόσιε συμβάσει θα συνεχίσουν να προκαλούν ένα επίπεδο λαθών πάνω από το όριο του 2%. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Άνερ είναι αν έχει εξετάσει η Επιτροπή πιθανές προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα λάθη που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και αν ναι, ποιες είναι αυτές. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ, Βλάσακ. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Άνερ για την ε, έκθεση που μόλις μας παρουσίασε. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω ε, υπάρχει και μια πρώτερη εργασία σε αυτή τη διαδικασία. Έγινε προσπάθεια απλούστευσης, έγινε προσπάθεια διόρθωσης και βεβαίως αυτή η διαδικασία προϋποθέτει κατάρτιση των υπηρεσιών, των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Με την εμπειρία λοιπόν και σιγά σιγά το ποσοστό σφάλματος έχει μειωθεί. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να, εστιαστώ, να εστιάσω την προσοχή μου ε, στην ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Επίσης, όταν γίνονται έλεγχοι που γίνονται βεβαίως σε πολλαπλά επίπεδα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ε, ερμηνείας των στοιχείων, ένα σύστημα ε, επικοινωνίας σχετικά με τα στοιχεία και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να μάθουν από τα λάθη των άλλων. Ε, γιατί με τον τρόπο αυτό, μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση. Επίσης, το κομμάτι των ε, ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων σε μερικά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ε, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες έτσι ώστε να γίνουν αλλαγές. Χρειαζόμαστε την ιδιωτική χρηματοδότηση. Επίσης, να ρωτήσω, προτείνετε κάποιες συστάσεις κατά αυτήν την έννοια. Πρόεδρος, κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Περέση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση ε, του κυρίου Άνε. Προφανώς ε, μία από τις μεγάλες ανησυχίες μας είναι να μειωθεί το ποσοστό των λαθών στη διαχείριση των ταμείων και ικανοποιούμε πάρα πολύ ακούγοντας ότι μειώθηκαν μέχρι και 50%. Ο κύριος Άνερ ανέφερε τη χώρα μου, την Ισπανία, ως μία από τις χώρες όπου γίνονται λάθη. Ακούγοντας αυτά που είπατε και από την ενημέρωση που μου δίνουν οι αυτόνομες περιφέρειες αλλά και η κεντρική κυβέρνηση στην Ισπανία, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε καθίσει να σκεφτείτε μήπως η μέθοδος που χρησιμοποιείτε, το έχετε αξιολογήσει, οδηγεί σε τέτοια σφάλματα διοικητικής φύσεως τα οποία αναφέρεται ως ελαφρά και ε, σοβαρά ε, σφάλματα. Μήπως είναι στη μέθοδο λοιπόν το σφάλμα ή είναι στην ουσία, στο περιεχόμενο, στο, στη δαπάνη την πραγματική. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς εσένα αγαπητέ Ντύρκ Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσύ προσωπικά έχετε καταβάλει πολλές προσπάθειες έτσι ώστε σε αυτές τις ε, ε, περιοχές σφάλματος ε, να βελτιωθεί η κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική. Όμως γνωρίζομαι ότι οι κανόνες στην υλοποίηση επιτόπου της περιφερειακής πολιτικής εξαρτάται ε, κατά πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την κατάσταση της τοπικής διοίκησης. Εάν το γενικό σύστημα στις χώρες μέλη παραμένει τοξικό ε, ή είναι μολυσμένο ας πούμε από αυτήν την ε, περιραίουσα ικανότητα, ε, τότε και στο μέλλον θα υπάρχουν τέτοια ασφάλματα. Και βεβαίω ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση, αλλά δεν ξέρω εάν οι ελπίδες αυτές είναι βάσιμε. Έχετε κάποια αποδεικτικά στοιχεία, έχετε μαρτυρίες ότι θα υπάρξει και διόρθωση από πλευράς των ε, τοπικών εθνικών ε, κυβερνήσεων. Θα υπάρξει βελτίωση της εφαρμογής ε, των κανόνων της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά βεβαίως δεν κάνουμε εμείς όλους τους ελέγχους δηλαδή δεν ελέγχονται τα πάντα, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, θεωρείτε ότι δημιουργούμε εδώ απλώς μια νησίδα τελειότητος ή ότι θα υπάρξει έτσι διάχυση των καλών αποτελεσμάτων σε όλες τις ε, πολιτικές. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Ναι κύριε Γκάιερ, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Ε, είναι θέμα αξιοπιστίας και ακεραιότητας όσο και εικόνας και κύρους των θεσμικών οργάνων μας. Ακριβώς ε, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας το κεφάλαιο και το θέμα και θα εξακολουθήσει να είναι και στο μέλλον. Κοιτάγοντας τα τελευταία χρόνια, κοιτάζοντας τα τελευταία χρόνια το 2006, 7 και 8, είχαμε εκτιμήσεις από το ελεγκτικό συνέδριο για τα σφάλματα της τάξης τουλάχιστον του 10 με 11%, το οποίο μειώθηκε στη συνέχεια το 9 σε τουλάχιστον 3%, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η μείωση. Αξιοσημείωτη αλλά θα περιμέναμε στο μέλλον έτσι μια διακύμανση μάλλον, ένα σκαμπανέβασμα γύρω από αυτό το ποσοστό, γιατί το 2009 δεν ήταν έτοιμα ακόμα όλα τα κράτη-μέλη, ούτε τα πιο δύσκολα προγράμματα και τα μεγαλύτερα. Πάντως, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το συνολικό ποσοστό σφαλμάτων. Και πιστεύω ακράδαντα, και επανέρχομαι στις ερωτήσεις που έγιναν για τις δυνατότητες, πιστεύω ακράδαντα λέγω ότι οι διοικητικέ ικανότητες στα κράτη-μέλη διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Να σας δώσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα σε εισαγωγικά βλέπετε τα κανονικά, τα αναμενόμενα προβλήματα σε κράτη-μέλη που είναι ακόμα στη φάση δημιουργίας δομών γενικά και διοίκησης. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τους βοηθούμε όσο γίνεται περισσότερο να φτιάξουν τη διοίκησή Παράδειγμα, ένα από τα προβλήματα που συναντήσαμε στη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου και της σημερινής είναι ότι είχαμε επενδύσει πολύ στην κατάρτιση συναδέλφων στα κράτη-μέλη. Είχαμε συναδέλφους πάρα πολύ καλά καταρτισμένους και παραμορφωμένους και τα Χριστούγεννα μας έστελαν ωραίες κάρτες ε, και μας έλεγαν μπορεί να σας εκπλήξει αλλά βρήκα θαυμάσια δουλειά σε μια ιδιωτική εταιρεία και τώρα δουλεύω ξέρω εγώ στην Price Waterhouse Cooper παράδειγμα ότι ωραία με καταρτήσατε και σηκώθηκα και έφυγα. Ε, τι θα κάνουμε για να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη όσο γίνεται να αυξήσουν τους μισθούς αλλά ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία ενδεχομένως να δημιουργήσουν δομές εκτός ε, ε, της κανονικής διοίκησης που έχουν αυτά τα στελέχη που είναι τόσο καλά καταρτισμένα και με τόσα πολλά προσόντα ώστε να παίρνουν και μισούς αντάξιους της δουλειά τους και να μη σηκώνονται να φεύγουν. Αυτή βέβαια είναι πυροσβεστική λύση και έκτακτες ανάγκη Γενικά δεν είναι σκόπιμο να ακολουθείτε. Άλλο παράδειγμα προσωπικό, έτσι, αλλά το λάβετε ως προσωπικό παράδειγμα, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια ενός ε, προγράμματος για τη μείωση των ε, δημοσίων υπηρεσιών του δημοσίου, οι χώρες ε, ρωτούν αν έχουν αρκετούς δημοσίους υπαλλήλους για να κάνουν τους ελέγχους. Ε, ήταν μια ιδιωτική εμπειρία, δεν θα σας αναφέρω την περίπτωση, αλλά Εκεί πολλές φορές είναι αξιοσημείωτα τα λάθη που γίνονται σε συχνότητα και μέσα μου αναρωτιέμαι μήπως επειδή μειώθηκαν τόσο πολύ υπάλληλοι. Όταν έχουμε δισεκατομμύρια δημοσίων πόρων να δαπανούμε χρειαζόμαστε μια πάρα πολύ γερή κρατική μηχανή, δυνατότητα διαχείρισης με σωστό τρόπο όλων αυτών των κονδυλίων. Εν μέρει έχουμε προβλήματα τα οποία δεν συνδέονται με τις δυνατότητες και τις ικανότητες, αλλά περισσότερο με συνταγματικές δυσκολίες σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ας πούμε υπάρχουν κράτη όπου υπάρχουν πολύ ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ κεντρικού κράτους, περιφερειακής διοίκησης και πολλές φορές έχουμε ανταγωνισμό για τις αρμοδιότητες. Ε, στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και καμιά φορά αυτό οδηγεί σε παράλυση, ξέρετε. Το έχουμε διαπιστώσει. Και μια που αναφέρεται και την Ισπανία, θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι αυτό δεν αφορά το σύνολο της Ισπανίας, αλλά ορισμένες αυτόνομες περιφέρειες θα μπορούσαμε να δούμε πού είναι τα προβλήματα. Και αυτό επίσης καταδεικνύει ότι δεν είναι αδύνατο να γίνει ε, σωστή διαχείριση των χρημάτων. Διορθώνονται αυτά. Λοιπόν, όταν διορθώνουμε ένα σφάλμα, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Όταν διορθώνουμε ένα σφάλμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βεβαίως και το καταχωρούμε και τη διόρθωση έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία και έχουμε πραγματικά ίχνος ε, καταγεγραμμένο της διόρθωσης. Το ελεκτικό συνέδριο τώρα έχει διαφορετική μέθοδο. Είναι φωτογραφική, ε, σας είπα, η παρατήρηση και κοιτάνε ανα πάσα στιγμή, σε μία στιγμή, κάθε ευρώ που έχει δαπανηθεί, ε, τι πιθανότητες έχει να ελεγχθεί. Και όταν τελειώσει η ετήσια εργασία προχωρούν στο επόμενο έτος με την ίδια μεθοδολογία η διόρθωση των σφαλμάτων που γίνεται εκ των υστέρων δεν εμφανίζεται πραγματικά στα στοιχεία τους. Ε, φέτος, ας πούμε στη Μάλτα ξέρω εγώ, μπορεί να έχουμε ένα σφάλμα το οποίο ανακαλύπτουμε, αλλά του χρόνου η Μάλτα να μην είναι καν στο δείγμα το οποίο ε, ελέγχεται και το γεγονός ότι διορθώθηκε το σφάλμα ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αποτυπώνεται με αυτή τη μέθοδο ε, στη μελέτη. Αν διακόπτουμε προγράμματα, στέλνουμε τη λειτουργία τους βεβαίως. Και συγκεκριμένα και ιδιαίτερα από την αρχή του έτους, του 2011. Διότι από την ανάλυση του 10 και μετά έχουμε πολλά χρήματα της περίοδου 2007-2013. Το καλοκαίρι ε, διέκοψα καμιά ογδονταριά προγράμματα στην περιφερειακή πολιτική. Ευτυχώς τα κράτη-μέλη και αρμόδιες αρχές αντέδρασαν αρκετά γρήγορα στις περισσότερες περιπτώσεις και από το Σεπτέμβριο επαναλήφθηκε η λειτουργία των προγραμμάτων αυτών και ε, έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όποτε υπάρχει αφιβολία, διακόπτεται το πρόγραμμα, να στέλνεται η ροή του και... Όταν δεν μπορούμε να διακόψουμε την εκταμείευση, την πληρωμή, θέλουμε αυτό που λέμε προειδοποιητικές επιστολές στις αρμόδιες αρχές για να πούμε ότι έχουμε βρει πρόβλημα και σε περίπτωση που υπήρχε εκταμίευση θα την είχαμε διακόψει. Αυτό ισχύει και για τους συναδέλφους στις διαχειριστικές αρχές που αντιδρούν λοιπόν στη συνέχεια και προσπαθούν να ξεπεράσουν τα σφάλματα. Συμφωνώ κύριε Βανιστερόι, τα κράτη-μέλη βεβαίως έχουν μεγάλη ευθύνη κατά αυτήν την έννοια και τολμώ να πω ότι ε, μέχρι ένα βαθμό ε, οι περισσότερες χώρες ε, γνωρίζουν, συνειδητοποιούν την ανάγκη αυτή και πραγματικά προσπαθούν να καλύψουν. Υπάρχει και ένα λιγότερο καλό νέο που είναι μια διαστροφή του ίδιου του συστήματος. Είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Από τη στιγμή που τα κοινοτικά χρήματα αυτή τη στιγμή ελέγχονται και εποπτεύονται με πιο αυστηρό τρόπο από ότι ε, από ο έλεγχος που γίνεται στο εθνικό κομμάτι της χρηματοδότησης υπάρχει μία τάση στα κράτη-μέλη όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, με, με, κάποια αμφιβολία, ας πούμε, τα κράτη-μέλη λένε καλύτερα να μην το κάνουμε με κοινοτικά χρήματα, με εθνικά χρήματα να γίνει. Αυτό ε, ίσως είναι καλύτερο για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και χειρότερο για τον τόπιο, τον εθνικό φορολογούμενο. Ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο ίδιος βαθμός πειθαρχίας παντού και σε κάθε μορφή χρηματοδότησης. αληθεύει ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα ε, έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα της επικάλυψης ελέγχων. Για την επόμενη περίοδο θα προσπαθήσουμε να ε, μην ελέγξουμε ε, ε, πολλά προγράμματα εκεί που όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Στις ε, χώρες μέλη που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου, και επειδή ενδεχομένως ο όγκος των προγραμμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, ε, τότε θα ε, διασφαλίσουμε να υπάρξει ένας έλεγχος ανά έτος. Και αν έχει γίνει έλεγχος από την Εθνική Αρχή, τότε δεν θα κάνουμε και εμείς. Ε, και το αντίστροφο, μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συμφωνίες με τις Εθνικές Αρχές. Και βεβαίως το ελεγκτικό συνέδριο είναι απολύτως ανεξάρτητο και βεβαίως πρέπει να είναι ανεξάρτητο λόγω της μεθοδολογίας που εφαρμόζει. Επίσης ε, υπάρχει πλήρης ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ ημών και των εθνικών αρχών. Πάντα όλοι έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει. για κάποια προγράμματα. θα ήθελα να συμφωνήσω και με τον κύριο Σταυρακάκη γιατί υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η προσοχή μας ε, επικεντρώθηκε πολύ περισσότερο, υπερβολικά ίσως, ε, στη, στο κατά δηλαδή στο κατά πόσον υπάρχουν ανομαλίες ή όχι ε, και παρατυπίες ή όχι το ζήτημα είναι τι γίνεται με το κάθε πρόγραμμα, δηλαδή μπορεί να έχει κανείς ένα εξαιρετικό πρόγραμμα όσον αφορά την έλλειψη παρατυπιών ε, και την ε, ε, υλοποίησή του, αλλά που να είναι ανώδυνο στο γενικότερο πλαίσιο. Και αναρωτιέται λοιπόν κανείς στο τέλος, ε, άξιζε τον κόπο να γίνουν όλα αυτά. Ναι, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται επί τόπου. Μερικές φορές δυστυχώς ε, στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής, μονάχα μετά από πάρα πολλά χρόνια μπορούμε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο επιτόπου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει μαζί με τα κράτη-μέλη να αναπτύξουμε μία μεθοδολογία βάσει της οποίας μπορούμε να έχουμε κάποιο, κάποια ένδειξη τουλάχιστον αποδοτικότητας ε, του προγράμματος επιτόπου. Και νομίζω ότι στη συζήτηση για την αξία ενός προγράμματος αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Κύριε Βλάζακ, ναι, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω απλούστευσης και ε, την προσπάθεια αυτή την καταβάλουμε. Όλοι μας λέμε ότι έστω και αν τώρα έχουμε μια καινούργια πρόταση, παρόλα αυτά ε, και για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα είμαστε ανοιχτοί έτσι ώστε οποτεδήποτε ε, έχουμε μία καλή ε, πρόταση απλούστευσης να την λάβουμε υπόψη μας. Πάντως ήδη για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχουν προβλεφθεί αρκετές απλουστεύσεις. Επίσης, στην επόμενη προγραμματική περίοδο ή μάλλον αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά την εθνική συγχρηματοδότηση, το τμήμα δηλαδή του εθνικό, θα υπάρξει η δυνατότητα χρηματοδότησης και από άλλες πηγές και όχι μονάχα δηλαδή από δημόσιο χρήμα, αλλά θα το ελέγξω και αν έχω κάνει λάθος θα μιλήσω μαζί σας προσωπικά. Η εντύπωσή μου είναι ότι πραγματικά έχουμε μπει σε ένα καλό δρόμο. Έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες από όλες τις πλευρές και οφείλω να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι όσον αφορά ε, τις ε, παρατυπίες ε, ελέγχονται όλο και περισσότερο και παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο αυτών των παρατυπιών, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η έλεγχη και ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα έρθω να σας μιλήσω θα έχω την δυνατότητα να πω περισσότερα γι' αυτό. Ε, ο στόχος σήμερα όμως ήταν πραγματικά να έχετε μια γενική πληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει όσον αφορά τα σφάλματα και τις παρατυπίες. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ, Dirk λέει η Πρόεδρος. Η νέα πολιτική ξέρουμε ότι θα είναι πιο προσανατολισμένη ε, προς τα καλά αποτελέσματα και η έλεγχη θα είναι πιο αποτελεσματική και σιγά σιγά θέλουμε αποτελεσματικότητα και της ίδιας της πολιτικής. Επομένως αξιολόγηση και στάθμιση της ίδιας της ε, ε, πολιτικής και όχι μονάχα των ε, σφαλμάτων και των ελέγχων. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι την πρωινή μας συνεδρία. Θα ξαναρχίσουμε στις 3 έτσι ώστε να έχουμε ε, παρουσία του ε, Επιτρόπου κυρίου Χάνα και της Πολωνικής Προεδρίας μια συνάντηση για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Σε ευχαριστώ πολύ.